Cher Chers collègues, bonjour. Καλημέρα. Si vous permettez, nous allons... Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα. Στις 10 ξεκινάμε ψηφοφορία σας, προειδοποιώ. Θα λάβατε την ημερήσια διάταξη. Έχετε μήπως προσθήκες, έχετε σχόλια όσον αφορά την πρόταση ημερήσιας διάταξης, όχι. Άρα μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο είναι η έγκριση των πρακτικών της ενηδριάσεως της 20 Ιανουαρίου 2015. Έχετε παρατηρήσεις. Προσθήκες δεν βλέπω να υπάρχουν. Θεωρώ ως εγκεκριμένα και τα πρακτικά στις ανακοινώσεις του Προέδρου τώρα. Μία μικρή αλλαγή. Λόγω της οθεσμίας καταθέσεως τροπολογιών στις δύο επιτροπές σήμερα το μεσημέρι άλλαξε η σειρά της ψηφοφορίας. Θα πρέπει ψηφίσουμε τις τροπολογίες που αφορούν την συμπερίληψη ισότητας των φύλων στην αρχή των ψηφοφοριών. Ε, το σημείο 8 και 9 θα ψηφιστούν πρώτα και μετά θα συνεχίσουμε με τα άλλα σημεία. Καλημέρα σας, Έτσι μπορούμε να διαβιβάσουμε τα ψηφίσματα στην Επιτροπή μας. Το τέταρτο σημείο αφορά τη συζήτησή μας για την κρίση του ιού έμπολα, διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις. Η συγγήτρια είναι η κυρία Τερέζα Χιμένες Μπεσέρι Μπάριο. Χαίρομαι που η Επιτροπή μας επεξεργάστηκε τη γνωμοδότηση αυτή ακόμα και αν η κρίση της έμπολα αποκλιμακώνεται ε, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Παρόλα αυτά θα πρέπει να προλάβουμε στο μέλλον κρίσης. Δίνω το λόγο αμέσως λοιπόν στην εισηγήτριά μας, την κυρία Χιμένεθ. Έχετε το λόγο. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση για την κρίση του έμπολα ήταν πάρα πολύ σημαντική για να δούμε πόσο, πόση σχέση έχει ε, το θέμα του ιού του έμπολα με τα δύο φύλλα γενικά. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες όπως ξέρουμε. Ο ρόλος τους ως γυναίκες σε κάποιες ε, χώρες της Αφρικής έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις, ε, κυρίως κοινωνικές στην κοινότητα στην οποία δουν. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες, οι οποίες λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα αυτό, γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους. Ο έμπολα, όπως είπε πάρα πολύ σωστά η Πρόεδρος, θα μπορούσε να είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί τα ναι, Συνεχίζει να είναι όμως προβληματική. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, συνεχίζει να δημιουργεί σεξουαλική βία, ιδιαίτερο στην Σιέρα Λεόνε. Και επηρεάζει κορίτσια τα οποία δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία και είναι αυτές οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες αυτό τον ΙΕ. το έπολα από το οποίο προσβλήθηκαν και η έκρηξη που δημιουργήθηκε τις έκανε πιο ευάλωτες σε, ε, και σε σεξουαλικά προβλήματα και σε επιθέσεις. Δύο, πάνω από 2.000 ε, προβλήματα έχουμε και τι ε, σημαίνει αύξηση του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύπλοκη και ανυπόφορη κατάσταση γυναίκες. Όλοι γνωρίζουμε ότι το νοσηλευτικό, παρανοσηλευτικό προσωπικό συνήθως είναι γυναίκες στα διάφορα νοσοκομεία. Ε, τα κορίτσια πρέπει να μένουν στο σπίτι, δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο αν έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό επιμένω να εγκρίνουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότης ώστε όλες οι γυναίκες την ε, Δυτική Αφρική και όλοι όσοι έχουν προσβληθεί από αυτό τον ιό να τύχουν υποστήριξη. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και προφορικές. Πρέπει να πω ότι συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά με τους υπολείπους συναδέλφους, του οποίους ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την εργασία που επιτέλεσε. Θα ήθελα και πάλι τελειώνοντας να σας ευχαριστήσω για την προσοχή με την οποία ασχοληθήκατε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ Τερέζα. Αρχίζει η συζήτηση. Η κυρία Χέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω για τη Μαρία Αριάννα που δεν μπορεί να παρίσταται. Θα διαβάσω. I would like to Λοιπόν, ευχαριστώ την εισηγήτρια την Τερέζα Χιμένεφ για τη δουλειά της και τις προτάσεις που έκανε συμβαστικές προτάσεις. Τη στηρίζω. Πολλές τροπολογίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Θεώρησα όμως ότι κάποιες ήταν εκτός πεδίου και θέματος και έτσι υποστηρίζω. Επιμένω ότι είναι αναγκαίο να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση των εγγύων γυναικών. Χρήζουν ιδιαίτερας μεταχειρήσεως. Και θα πρέπει να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη με εκείνους που τις φροντίζουν και ελπίζω ότι οι σχετικές τροπολογίες θα στηριχθούν. Αυτά είπε η Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ πολύ. Άννα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Βερονίκ Λορέντσο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευράς μας πρέπει να πω την άκουσε ευπρόσδεκτη. Η έκφραση ανησυχίας του κειμένου και συμφωνούμε η έμπολα εξελισσόταν συνεχώς και έπληξε ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα κορίτσια σαν εκπαιδεύτριες, σαν άνθρωποι που παρήχαν περίθαλψη, σαν μέλη σαν οικονομικοί συντελεστές ο ακριβής αντίκτυπος της επιδημίας στις γυναίκες και τα κορίτσια είναι άγνωστος ακόμα. Ξέρουμε ότι ήταν πολύ σοβαρός ο αντίκτυπος και ξέρουμε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες που στηρίζει συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επλήγησαν, κυρίως έκλεισαν και η συνηθισμένη παροχή περίθαλψης μειώθηκε. Άρα πολλές γυναίκες δεν θα είχαν πρόσβαση σε προγεννητική φροντίδα ή βοήθεια κατά τη της γένας. Ξέρετε ότι θέλει να βοηθά τις χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία και να κερδίζουμε έτσι. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια, που δεν έχουν πρόσβαση σε υγεία και παιδεία και υποφέρουν από ανισότητες και από την έλλειψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό θα εφαρμοστεί και στην περίοδο μετά την επιδημία της έμπολα και την περίοδο αποκατάστασης. Ο σχεδιασμός των έργων που αφορά τα στήματα υγείας πρέπει να οδηγήσει ενίσχυση αυτών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την ισότητα των φύλων. Να καλύψουμε πολλές πτυχές συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων κατεβλήθησαν πολυσχηδείς προσπάθειες από την ΕΚΟ και από εμά να μειώσουμε τα συμπτώματα, τα κρούσματα ε, και έχουμε φτάσει σχεδόν στο μηδέν. Το τελευταίο 10% είναι το δυσχερέστερο και χρειαζόμαστε μεγαλύτερες προσπάθειες ούτω ώστε να διακοπεί η μετάδοση και έτσι να μην έχουμε απώλειες ζώων. Διαπιστώνουμε ότι η επιδημία της έμπολα τόνισε την ανάγκη ισχυρών συστημάτων υγείας, της εκπαίδευσης, της διακυβέρνησης και είναι πτυχές που λαμβάνουμε υπόψη στις αξιολογήσεις για την ανάκαμψη από την έμπολα που διενεργούνται από τον ΟΗΕ μαζί με μας και την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους, ούτως ώστε να παραχθούν εθνικά σχέδια που θα εδράζονται επιεθνικής συμμετοχής και δυναμικού. Θα δώσουμε προσοχή σε στοιχεία με βάση το φύλλο και ποια είναι τα βασικά αιτήματα των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών. Ξεκινήσαμε σαν ΤΕΦΚΟ την ανάλυση των συστημάτων υγείας. Είχαμε ξεκινήσει ήδη κατά την ε, περίοδο εκτάκτου ανάγκης εστιαστήκαμε επί δύο πυλώνων, ενίσχυση των συστημάτων υγείας και ετοιμότητα των περιοχών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν συνεργασία μαζί σας, με τις επιτροπές σας, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε τα μαθήματα που πήραμε και να εφαρμόσουμε τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της βοηθείας. Και θέλουμε αυτά τα σχέδια να τα στερνίζονται οι κυβερνήσεις οι συνεργαζόμενες με εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λορέντσο. Ευχαριστώ λοιπόν. Είχαμε ελπίσει ότι θα επιτυχάναμε να ανακόψουμε την ε, διάδοση του ιού έμπολα. Διότι τελικώς κινδύνευε ολόκληρος ο κόσμος. Στη ρίζα του κακού αυτού βρισκόταν και έλλειψη των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων, ανεπαρκές προσωπικό και ούτε καθεξής προβλήματα και βεβαίως υποδομών προβλήματα τα οποία υπήρχαν στις χώρες αυτές ενδυμικά και πριν από την ε, έκρηξη της ε, επιδημίας. Και αυτό επέτρεψε, ή αυτά επέτρεψαν την ταχύτατη διάδοση του ιού. Η κατάσταση στις χώρες που έχουν πληγεί δεν καθιστά δυνατό να ανακοπεί τελείω η διάδοση του ιού. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Σε φτωχές χώρες είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαρκής υγειονομική υποδομή και εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτά έχουν μεγάλη σημασία. τα καλύτερα προληπτικά μέτρα είναι μια γερή υγειονομική υποδομή. Τούτη τη φορά ήταν βέβαια ο ιός του έμπολα. Υπάρχουν όμως κι άλλα. Ελονοσία, φυματίωση. Από αυτές τις βαριές αρρώστιες πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Ας μην το λησμονούμε αυτό. Όλοι εμείς που ασχολούμεθα με την πολιτική αναπτύξεως θα παρακαλέσω τώρα την κυρία εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Τέρεζα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που θα ήθελα να κάνω ευχαριστώ τους συναδέλφους και να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις που έκανε και η Επιτροπή. Τελικά έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα δημόσιας υγείας και πώς θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε κάτι για να βελτιωθεί η δημόσια υγεία στις χώρες αυτές. Η Επιτροπή Ανάπτυξη επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και μετά από συναντήσεις με υπεύθυνους από τις περιοχές αυτές θα πρέπει να μας πούνε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που διαθέτουμε ώστε και στα νοσοκομεία, κυρίως σε μικρά νοσοκομεία στην Ήπεθρο μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα η ασθένεια αυτή διότι μεταδίδεται πολύ εύκολα. Εμείς ε, στέλνουμε οικονομική βοήθεια, αλλά θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουν καλύτερα. Κυρίως ανέφερα το πρόβλημα το οποίο είναι πιο οξύ για τις γυναίκες, για τις έγκυες γυναίκες, ε, όπως αναφέρθηκε και από την Μαρία Ρένα. Πρόκειται για θέμα υγείας, δημόσιας υγείας, που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια, τις γυναίκες που παραδοσιακά ε, βρίσκονται πιο κοντά στους ασθενείς, τους οποίους φροντίζουν. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστώ πολύ. Προστεμία κατάθεσης τροπολογιών ήταν η 6η Φεβρουαρίου το μεσημέρι κατατέθηκαν 73 ε, τροπολογίες και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 10. Σας ευχαριστώ. Περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015. Η συγγήτρια, η συνάδελφος Μαρία Νόιχλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την προσοχή που χάρισατε στο θέμα μου στρατηγική για την ισότητα των γυναικών μετά το 2015. Η έκθεσή μου είναι έτοιμη, είναι η πρώτη μου έκθεση ως Ευρωβουλευτού. Η σύνταξη της έκθεσης ήταν υπόθεση που μου πρόσφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση. Έχουν γίνει συζητήσεις και εδώ στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Βεβαίως έγινε πολύ καλή συνεργασία και με τις κοιόδης συγγήτριες. Ευχαριστώ όλα τα όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Έχω να πω κάτι και για τις ομάδες της κοινωνίας των ε, πολιτών ή τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δηλαδή οι οποίες από την αρχή <clears throat> κράτησαν επαφή μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σημαντική της βοήθεια. Εγώ έχω χωρίσει την έκθεσή μου επίτηδες έτσι ώστε να δείξω καθαρά ότι δίνουμε σημασία σε όλα τα κεφάλαια εντό εισαγωγικών εκείνα τη ζωή τη γυναίκα όπου ενδέχεται αυτή να υποστεί διακριτική μεταχείριση. Δεν έχω τηρήσει απόλυτα την ταξινόμηση που είχε ε, κάνει η προηγούμενη ε, έκθεση. Έτσι έχω λοιπόν ένα πρώτο θέμα γενικές συστάσεις μετά προχωρώ βία κατά των γυναικών, που νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και το υπαριθμόν ένα θέμα, έτσι με αυτό αρχίζει την ουσία η έκθεση. Προχωρώ στο άλλο θέμα εργασία και χρόνος, μετά δημιουργικές ικανότητες, οικονομικά μέσα, υγεία, γνώση, εκπαίδευση, μέσα ενημέρωσης, η παγκόσμια οπτική και τέλος οι θεσμικοί μηχανισμοί. Μιλώντας σήμερα για ισότητα, έχει κανείς την αίσθηση ότι Υπάρχουν ποικίλε στάσει απέναντι στην ισότητα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι ήδη έχουμε πετύχει την ισότητα. Άλλοι πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμα απόσταση. Πάλι άλλοι, οι άλλε, λένε ότι είναι υπερβολικά δαπανηρό το να πετύχει κανεί την ισότητα, ιδίω σε περίοδους κρίσεων. Και τέλο υπάρχουν και εκείνε που πιστεύουν ότι η ισότητα είναι σημαντική και πρέπει να προωθηθεί. Ο δρόμο βέβαια μέχρι την εξασφάλιση της ισότητας είναι μακρύ. Η gender equality έχουμε φαίνεται πετύχει 54 από συνολικά 100 ε, δυνατά σημεία. Ενδεχόμενα δηλαδή με την έννοια αυτή. Όμως η ισότητα θα αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα κοινωνικά και οικονομικά για ολόκληρη την κοινωνία και για την ανδρική πλευρά. Πρόκειται για ανθρώπινο δικαίωμα. Αλλά δεν είναι τελικά το εάν θα τα πάει καλύτερη, καλύτερα η οικονομία ή θα τα πάει καλύτερα ο Α ή Β κράτος, αλλά είναι ανθρώπινο δικαίωμα η απόλυτα ισότιμη μεταχείριση. Τα επόμενα πέντε χρόνια λοιπόν πρέπει επιτέλους να αναλυθούν κάποιες δράσεις. Βασικό στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να είναι μια συνεκτική στρατηγική. Στρατηγική όμως σημαίνει όχι μόνο να διαπιστώσει κανείς που υπάρχουν ελλείψει, στρατηγική σημαίνει και ενθάρρυνση, προτροπές για ανάληψη δράσεων, για την αντιμετώπιση όλων των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα τονίσω τώρα ορισμένου επιμέρους τομείς. Μία οδηγία η οποία προβλέπει ένα σύστημα καταγραφής προσωπικών δεδομένων και βεβαίως και για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Τέτοια οδηγία είναι αναγκαία και απαραίτητη. Η κύρωση τη συνθήκη τη Ισταμπούλ για την αντιμετώπιση τη βία κατά των γυναικών. Πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω και από όλε τι χώρε μέλη. Σε μικρή αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΦΕΜ ήμουν παρούσα στην Ρήγα. Η Λετωνία λοιπόν μετά από κατ' επανάληψη υποβολή ερωτήσεων μας είπε ότι το 2016 θα κυρώσει την συνθήκη της ε, Ισταμπούλ. Το έτος του 2016 θα λάβει την ονομασία έτος της καταπολέμησης της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα να μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ευρώπη το 2016. Άλλο σημαντικό θέμα, και βεβαίως γνωρίζετε τη σχετική συζήτηση, είναι και η ψήφιση της οδηγίας για τη μητρότητα πρόκειται για μια κρίσιμη φάση στη ζωή της γυναίκας όπου χρειάζεται η γυναίκα ιδιαίτερη προστασία. Παρόλο τον οικογενειακό σχεδιασμό, παρά το ότι δημιουργείται μια οικογένεια, πρέπει να εξασφαλιστεί και η δυνατότητα συνδυασμού της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Και πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο και οι άνδρες. Δεν θέλουμε μονάχα να πάρουμε εμεί οι γυναίκες, αλλά θέλουμε και να δώσουμε. Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα στους άνδρες να ασχοληθούν με την οικογένεια και με τα οικιακά. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, βεβαίως και δεν μπορεί να γίνει αυτό νομικά επιβεβλημένο καθήκον. Διάβασα σε μια γερμανική εφημερίδα ότι πάμε εδώ λέει να επιβάλλουμε καθήκοντα στους άνδρες. Όχι, δεν είναι αυτό το νόημα. Η οικογενειακή δομή όμως πρέπει να προβλέπει ότι συμμετέχει και ο άνδρας. Η ψήφιση της οδηγίας για ισορροπημένη ε, εκπροσώπηση των δύο φίλων σε εποπτικά συμβούλια. Και αυτό είναι ένα κέριο βήμα. Θέλουμε επίσης να ληφθούν μέτρα για διαφανέστερη διαμόρφωση των αμοιβών. Να γνωρίζουν όλοι και όλες ποιος κερδίζει πόσα και για ποιο λόγο. Σε ορισμένε χώρε τα πράγματα αυτά καλύπτονται από ένα πέπλο αδιαφάνεια. Σαν να είναι απόρριτα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτή η μεγάλη απόσταση των αμοιβών που εξακολουθεί να υπάρχει πρέπει να μειωθεί και πρέπει να εξαλειφθεί. Επίσης, οι υπηρεσίες για την αναπαραγωγική υγεία. Επίσης πολύ σημαντικός τομέας θέλουμε ασφαλείς νόμιμες δυνατότητες και πρόληψης της εγκυμοσύνης και άμβλωσης. Σημαντικό αυτό επίσης έχει ε, απασχολήσει πολύ και τον τύπο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο να προσελκύσουμε τις γυναίκες οι οποίες μπορεί να θέλουν το παιδί να προχωρήσουν σε άμβλωση. Καθόλου μάλιστα. Εάν μια γυναίκα ωστόσο αποφασίσει ότι επιθυμεί να προχωρήσει σε άμβλωση, αυτό είναι δική της ατομική απόφαση. Τότε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η γυναίκα αυτή δεν προχωρεί στην άμβλωση αυτή χωρίς ιατρική παρακολούθηση, χωρίς υποστήριξη. Όλες γνωρίζουμε από τις χώρες μέλη μας, δεν είναι άλλωστε και τόσο παλιά υπόθεση αυτή, ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πεθαίνουν από αιμορραγία στη διάρκεια της άμβλωσης. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν να προωθήσουμε την ιδέα της άμβλωσης, απλά όταν πρόκειται να γίνει η άμβλωση να γίνεται με σωστό τρόπο. Επίσης η διατήρηση της ισότητας των φύλων πρέπει να είναι κριτήριο και για όλα τα προγράμματα έρευνας, για, γειτονική, για πολιτική γειτονία δηλαδή και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά. Και εκεί λοιπόν πρέπει να διαφυλάσσονται απαραίτητο τα δικαιώματα των γυναικών και να περιλαμβάνονται σε όλες αυτές τις ε, συμφωνίες και συνθήκες. Το ίδιο για το άσυλο και την πολιτική μετανάστευση. Έκανα την προσπάθεια λοιπόν με τα λόγια αυτά να σας εξηγήσω ορισμένα βασικά σημεία της έκθεσης που ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμη. Εγώ δεν κατόρθωσα να περιλάβω όλα τα θέματα που με ενδιαφέρουν τις λίγες αυτές σελίδες που ε, έχω στη διάθεσή μου. Σας παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε την έκθεση, να μου στείλετε τις τροπολογίες σας, γιατί θέλω με κοινή προσπάθεια να τις περιλάβουμε και να φτιάξουμε τελικά ένα έγγραφο το οποίο να εξυπηρετεί τις γυναίκες στην Ευρώπη αλλά βέβαια και τους άντρες και να επιτρέψει σε όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Μέχρι τις 5 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τροπολογίες και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα προκύψει. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, εισηγήτρια, κυρία Νόιχελ, για την ε, ενδιαφέρουσα αυτή τοποθέτηση. Ε, η κυρία Πέτη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα θα μιλήσω εν ονόμα της κυρία Κάρτερς που λυπάται πολύ που δεν μπορούσε να παραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση αλλά μου ζήτησε παρόλα αυτά να διαβιβάσω εν ονόματί της κάποιες σκέψεις. Η κυρία Γκάλπερς δέχτηκε θετικά το έργο της εισηγήτριας όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το 2015 που είναι αποφασιστική σημασία για περαιτέρω αποτελέσματα στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Πρέπει να είναι ένα στόχο σημαντικότατος για όλους μας, μια προτεραιότητα διότι ε, παράγει θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε στο μέλλον όπως κατά παρελθόν να κινηθούμε στον τομέα και η κυρία Γκάλπελτς πιστεύει ότι αυτή η έκθεση μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε επικοδημητικό διάλογο με όλους τους συμμετέχοντες στην όλη διαδικασία. Η κυρία Γκάλπελτς ενθαρρύνει την εισηγήτρια να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό όπως μέχρι τώρα στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα ποιοι ήταν οι στόχοι που επιτέχθηκαν στο παρελθόν και τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κυρίως όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Έχουμε ήδη ένα πακέτο για τα θύματα, αποτελεί τμήμα ενός ευρυτέρου πακέτου νομοθετικού για μας πρέπει να πούμε ότι ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου για την εναρμόνιση της νομοθεσίας στα διάφορα κράτη-μέλη και το πώς εφαρμόζεται. Η κύρωση της συμβάσεως της Κωνσταντινούπολης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών είναι μεγάλη σημασία. Όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για τη μητρική άδεια που μπλοκαρίστηκε το 2010 στην πρώτη ανάγνωση δυστυχώς. Είναι απίθανο το Συμβούλιο να μπορέσει να προχωρήσει πάνω σε αυτό. Εν γέννη, η θέση της κυρίας Γκάλπελς είναι ότι όλα τα επιχειρήματα που αφορούν, όλα τα θέματα μάλλον που αφορούν την επικουρικότητα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των 100 μελών. Η κυρία Γκάλπελ θέλει να συνεχιστεί η συνεργασία με την εισηγήτρια και του κοιόδης εισηγητέ πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα. Αυτή η έκθεση είχε σαν βασική ιδέα να οδηγήσει σε μια ανάπτυξη μια στρατηγικής για την ισότητα καθώς και την καταπολέμηση εμπορίου ανθρώπων. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία με τα οποία ίσως να μην συμφωνούμε όπως η πρόθεση της άμβλωσης και η ισοτιμία όσον αφορά τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων θα πρέπει και τα δύο φύλλα να συνεργάζονται, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και φυσικές διαφορές μεταξύ των φύλων. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι η κατάσταση των νέων μητέρων ε, θα βελτιωθεί. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η μητρότητα και η πατρότητα θα υποστηρίζονται. Η καταπολέμηση της βίας έχει μεγάλη σημασία και αυτή. Η βία όμως απαγορεύεται αυτή καθεαυτή σε όλα τα κράτη-μέλη. Διαφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε την έγκριση της συμβάσεως της Κωνσταντινούπολης. Η Πολωνία από την πλευρά της δεν πιστεύει ότι θεσπίζονται νέες διατάξεις από τη σύμβαση. Είναι ένα ιδεολογικό κείμενο όσον αφορά το περιεχόμενό του. Διότι ο βασικός λόγος για την διάπραξη βίας κατά των γυναικών είναι το ενόπνευμα, κατάλληλος ενόπνευματος, καθώς και το πώς προβάλλεται η εικόνα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Και είναι εσφαλμένο πιστεύω να θεωρείτε ότι η βία μπορεί να προέρχεται από θρησκευτικού λόγους Φερρυπίν. Διαβάζουμε επίση ότι κάθε δεύτερη γυναίκα είναι θύμα ε, βίας. Αυτά τα στοιχεία διορωτώμα από πού προέρχονται. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι αξιόπιστα. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013 αναφέρει σαφώς ότι η άμβλωση και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρόσφατα. Η νέα στρατηγική για την ισότητα δεν περιέχει τέτοιες πτυχές. Πιστεύω ότι δικό μας καθήκον είναι η βελτίωση της θέσεως των γυναικών και όχι η πρόθεση της άμβλωσης, διότι η γυναίκα είναι επίσης θύμα ε, της άμβλωσης. Δεν είναι δικαίωμα κανενός. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν τμήμα της υγείας ούτε του οικογενειακού σχεδιασμού. Η αδίποτε άμβλωση είναι επικίνδυνη για τη ζωή και την υγεία της γυναίκας. Καθήκον μας είναι να προστατεύουμε τη γυναίκα και το παιδί και στην προγενετική φάση καλή ε, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι η σωστή προσέγγιση. Χρειαζόμαστε καλά καταρτισμένο, εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό. Τα στερεότυπα όσον αφορά τους ρόλους ανδρών και γυναικών ευράζονται σε πολιτισμικά στοιχεία και στην παράδοση. Δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσει τα παραδοσιακά στερεότυπα και τους ρόλους κυρίως εμείς σαν κοινωνία που ε, επιδιώκουμε την ευτυχία και τα υλικά αγαθά ε, πολύ συχνά υποτιμούμε το ρόλο της μητέρας. Είναι σαφές ότι θα είχε νόημα αν συμμετείχαν περισσότερες γυναίκες στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Δεν είναι ρόλος όμως του Κοινοβουλίου να ανακατευθεί ε, στις νομοθεσίες των κρατών μελών και να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δικούς της κανονισμούς. Ε, δεν χρειαζόμαστε νέους νόμους που θα καθιστούν τις γυναίκες ε, να βρίσκονται μάλλον να προωθούν τις γυναίκες σε καλύτερη θέση στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η κυρία Αγγελικά Μλινάρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και σας κυρία Νόιχλ. Σας συγχαίρω άλλωστε, ρητά, για την εξαίρετη έκθεσή σας, καθώς και για το ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας. Είμαι ευτυχής που η έκθεσή σας επιλέγει μια ολιστική προσέγγιση. Κάτι το οποίο ταιριάζει πολύ και στη δική μας ιδέα. Και ευχαριστώ επίσης που περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στη γονιμότητα ως θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, έχω δύο ή τρεις συγκεκριμένες παρακλήσεις. Στην παράγραφο 5, όπου μιλείτε για τα διάφορα στοιχεία για κάθε φύλλο. να λάβετε υπόψη το Ινστιτούτο τη ισότητα. Υπάρχει. Υπάρχουν Ινστιτούτα δηλαδή τα οποία έχουν συλλέξει σχετικά στοιχεία. Άρα δεν χρειάζεται να επινοήσουμε εκ νέου τον τροχό. Υπάρχουν τα πράγματα αυτά. Στη δε παράγραφο 6 θα παρακαλέσω να λάβετε υπόψη και το νομοθετικό πρόγραμμα βέβαια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετικό πρόγραμμα συγκεκριμένο, διότι αλλιώ τα πράγματα μένουν στα λόγια. Τώρα, για το κεφάλαιο οικονομικά μέσα. Εκεί προτείνω να λάβουμε υπόψη το gender gap, δηλαδή αυτό το κενό, το χάσμα μεταξύ των φύλων, στις συντάξεις. Και τέλος, μια πραγματική παράκληση. Είπατε αρχικά ότι η προθεσμία κατάθεσης σχολείων δηλαδή τροπολογιών, είναι η 5η Μαρτίου. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σύντομο δηλαδή, το χρονικό διάστημα. Γνωρίζω ότι η Κομισιόν πάει να φτιάξει μια πολύ ευρεία πρωτοβουλία. Σα παρακαλώ, αν είναι δυνατό, να παρατείνετε κατά τουλάχιστον μία εβδομάδα την προθεσμία αυτή. Η κομισιον παει να φτιαξει μια πολυ ευρια πρωτοβουλια σα παρακαλω αν ειναι δυνατο να παρατεινετε κατα τουλαχιστον μια εβδομαδα την προθεσμια αυτη η προεδρος σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, η κυρία Μορβάη.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 If today there Α, ζητώ συγγνώμη, δεν υπάρχει σήμερα ουγγρική μετάφραση. Θα τα πω στα αγγλικά. Εκφράζω την έκπληξή μου, ωστόσο, διότι συνήθω έχουμε ουγγρική μετάφραση. Παρακαλώ να εξετάσει η γραμματεία γιατί και να προβληθεί για την επόμενη φορά. Θα τα πω στα αγγλικά, λοιπόν. Να λοιπόν άλλο ένα έγγραφο όπου η άμβλωση παίζει ένα κεντρικό ρόλο και ορισμένες από τις παρατηρήσεις μου θα στρέφονται γύρω από μια, πώς να πω, ένα νέο σχεδιασμό της προσέγγισής μας γύρω από την άμβλωση ως φεμινίστριες ή τέλος πάντων ως υπέρ των γυναικών γενικότερα. Και πρώτα θεωρούμε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φαίνεται λέγω, την άμβλωση σαν κάτι το προοδευτικό, σύγχρονο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια μετατόπιση της νοοτροπίας ως ότι η άμβλωση είναι κάτι το αρχαϊκό. Εύχομαι στο μέλλον η άμβλωση να είναι μια κακιά ανάμνηση του παρελθόντος. Όταν δηλαδή οι γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να περάσουν μέσα από αυτή την οδυνηρή διαδικασία, οδυνηρή και ψυχολογικά και σωματικά και πνευματικά, διανοητικά. Όταν μιλούμε για τον σύγχρονο κόσμο, έχουμε και βεβαίως όλα σε αυτές τις διαγνωστικές δυνατότητες μέσω των οποίων τώρα γνωρίζουμε όλο και περισσότερα σχετικά με το έμβριο και την ανάπτυξή του και όπως λοιπόν ε, καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερο είναι όλο και πιο αρνητικό να αρνηθούμε ως φεμινίστες και γυναίκες τέλος πάντων πολιτικοί που ε, επιδιώκουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι όλο και πιο δύσκολο να αρνηθούμε ότι ότι και διανοητικά και σωματικά και ψυχολογικά είναι βαριά και οδυνηρή υπόθεση να καταστρέψουμε αυτό το πλασματάκι. Ας μην το αρνηθούμε αυτό πια, λέγοντας ότι εάν είμαι φεμινίστρια και προοδευτική κτλ. Το απορρίπτω αυτό ως θέμα. Θα ήμουν ευγνώμων λοιπόν αν μπορέσετε στο κείμενό σας να δείξετε αυτή τη μετακίνηση προσεγγίσεων στο έγγραφό σας και να διατυπώσετε το θέμα κάπως ένα όραμα δηλαδή ότι προσβλέπουμε σε ένα κόσμο όπου δεν θα υπάρχει ανάγκη πια να γίνονται αμβλώσεις. Γιατί, γιατί οι γυναίκες θα έχουν απόλυτο έλεγχο του σώματός των, γιατί θα αλλάξουν οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα είναι και φυσικό πλέον για τους άνδρες να αισθάνονται την ευθύνη για τις ε, συντρόφους τους, είτε πρόκειται για μια συνάντηση μιας βραδιάς ή αν πρόκειται και για ένα γάμο. Θα είναι απόλυτα φυσικό δηλαδή για τους άνδρες να εξασφαλίζουν ότι αν έχουν ερωτικές ερωτικέ σχέσει μια γυναίκα να μην την καταστήσουν έγκυο παρά την θέλησή τη, γιατί θα είναι πλέον θεμελιώδε ηθικό θέμα και για του ίδιου του άνδρες. Να αρχίσουμε λοιπόν να βάζουμε τα πράγματα αυτά μέσα στι εκθέσει μα. Όχι να συνεχίζουμε και να συνεχίζουμε επί δεκαετίε και να λέμε Α, άμβλωση είναι δικαίωμα των γυναικών και τμήμα τη ελευθερία του. Όχι, α αρχίσουμε να βάζουμε προτεραιότητα στα θέματα εκείνα που θα στηρίξουν τις γυναίκες στην πραγματική ζωή τους. Δηλαδή πρόληψη βεβαίως, πρόληψη της ανάγκης των αμβλώσεων με σύγχρονους ασφαλείς τρόπους οικογενειακού σχεδιασμού όπου οι άνδρες θα παίζουν το ρόλο του εταίρου και το άλλο, δεν ξέρω αν είναι και θέμα μετάφρασης ενδεχόμενα ή εγώ τέλος πάντων να μην κατανόησα καλά, αλλά μου φάνηκε ότι είπατε ότι, ότι οι γυναίκες εάν επιλέξουν την άμβλωση θα πρέπει να υποστηρίζονται στην επιλογή τους αυτή. Αν όμως πρόκειται για ένα, μια εγκυμοσύνη που δεν την έχουν σχεδιάσει και δεν θέλουν να προχωρήσουν στην άμβλωση αλλά προτιμήσουν να κρατήσουν το παιδί θα πρέπει να υποστηριχθούν και σε αυτή την δυνατότητα τότε. Συγγνώμη, μιλώ ακόμα στην εισηγήτρια, παρακαλώ μην την απασχολείτε. Ας φροντίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρχει ε, θεσμική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, γυναίκα προς γυναίκα και ψυχολογική και για κάλυψη των κοινωνικών της αναγκών και για κάλυψη των πνευματικών της αναγκών για γυναίκες οι οποίες δεν σχεδιάζουν ή δεν σχεδίαζαν αρχικά να μείνουν έγκυοι αλλά αποφασίζουν τελικά να κρατήσουν το περι Αυτά τα πράγματα εγώ τα θεωρώ πραγματικά σύγχρονα και προοδευτικά. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τα σκεφτείτε αυτά τα πράγματα και να τα περιλάβετε στο έγγραφό σας. Και επίσης να βρούμε και κάποια πράγματα ακόμα. Σήμερα, το 2015, γυναίκες και άμπλωση. Να μάθουμε ακόμη, να δείξουμε δηλαδή, γιατί άραγε οι γυναίκες χρειάζονται ακόμα τις αμβλώσεις ενώ έχουμε τόσο πολύ περισσότερο έλεγχο για, πάνω στα σώματά μας και τις ζωές μας, γιατί χρειαζόμαστε ακόμα ως γυναίκες την άμβλωση. Και επίσης ποια μορφή μπορεί να λαμβάνει η θεσμική στήριξη και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των γυναικών που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση όταν έχουν δηλαδή πλέον μια μη σχεδιασμένη ή μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. να ρωτήσουμε τις ίδιες τις γυναίκες να μην τους επιβάλλουμε μια συγκεκριμένη ιδεολογία χωρίς να ρωτήσουμε καν την άποψή τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τι κάνουν με τη ζωή τους και με τη σεξουαλικότητα Σας ευχαριστώ πολύ Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. κυρία Μορβάη Έχουμε ακόμη μόνο 10 λεπτά στη διαθέσή μας πριν από την ψηφοφορία. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή, από την κυρία Βίκερμαν, να μας πει ποια είναι η θέση της. Πέντε λεπτά δίνω λοιπόν στην Επιτροπή και πέντε λεπτά για τα συμπεράσματα στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νόησουλ για την πολύ πλήρη έκθεσή της και για τις διαβουλεύσεις τις οποίες κάνατε με όλους τους ενδιαφερομένους και τις ΜΚΙΟ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να πω ότι δεδομένου ότι η παρούσα στρατηγική ολοκληρώνεται το 2015, σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι μελλοντικέ προκλήσεις για να προωθηθεί σε ό,τι μεταξύ ανδρών και γυναικών τα επόμενα χρόνια και θα θέλαμε να ακολουθήσουμε μία διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους. Μπορώ να σας ενημερώσω για το εξής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που αποτελείται από ΜΚΟ, ε, κοινωνικού εταίρου και προσώπους καταμένων ήδη έχει υιοθετήσει γνωμοδότηση για προτεραιότητες και προκλήσεις για το θέμα αυτό για τα επόμενα χρόνια και η γνωμοδότηση αυτή, η έκθεση αυτή θα αποτελέσει την ε, δεύτερη πολύ σημαντική βάση συζήτησης για την επόμενη χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιεύσουμε την ετήσια έκθεση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών το 2014. Πρόκειται για την ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφεται η πρόοδος και η εφαρμογή της παρούσης στρατηγικής και τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στα πλαίσια του Ευρωβαρομέτρου. Πρόκειται λοιπόν για στοιχεία και δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε την περαιτέρω σκέψη μας. Υπάρχουν και προτεραιότητες και άλλε παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση που μας αφορούν. Βεβαίω θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να πληρωθούν τα κενά που υπάρχουν σε θέματα λήψη αποφάσεων, συνταξιδότησης και και πιστεύουμε ότι η εκθεσή είναι μία προτεραιότητα και θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να υπάρχει και συγκερασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και να προωθεί ισότητα μεταξύ των διευθύνων. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω βήματα για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών και πιστεύω ότι η σχετική σύμβαση θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό το θέμα. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπίκερμαν για τα συμπεράσματα η κυρία Νόιχελ. Πρώτα επιθυμώ να σας ευχαριστήσω όλες για τις ε, ενδιαφέρουσες προτάσεις. Προσπάθησα να τις σημειώσω όλες, να περιλάβω στην έκθεσή μου τα θέματα που θέσατε, δεν θα αφήσω ούτε ένα απ' έξω. Παρακαλώ μόνο συντάξτε τροπολογίες να ολοκληρωθεί με τον τρόπο αυτό η έκθεση. Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νόιχελ. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η προθεσμία για τις ε, κατάθεση τροπολογιών. Παρατάθηκε η προθεσμία αυτή έως τις 10 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Παράταση λοιπόν της προθεσμίας έχει ως τις 5 αλλά ως τις 10 Μαρτίου. Και μετά προβλέπεται η εξέτασή του στην συνεδρίαση της 21ης Τρίτου και στην ψηφοφορία στις 5 και 6 Μαΐου και στην ε, ε, εξέταση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ιουνίου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία στον αφορά τις τελευταίες ημερομηνίες. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Όπως ε, είπα και στην αρχή της συνεδρίασης, αρχίζουμε με τα ψήφιση των ε, εκθέσεων 8 και 9. Το gender mainstreaming πρώτα απ' όλα. όλα θα ψηφίσουμε την έκθεση της, της τη στην ίντα. Θα προτείνω να ψηφίσουμε το θέμα αυτό on block. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνούμε στην επόμενο θέμα. Green Grown Opportunity for SMEs. Τροπολογία 5. Υπέρ. Yes, please. Uh, What are we voting? We didn't... Τι ακριβώς ψηφίζουμε. Δεν καταλάβαμε, λέει ο Είπα στην αρχή της συνεδρίασης ότι ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα τα σημεία 8 και 9. Έκθεση 9. Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. man Pour. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει ένα τρίτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος πρώτα απ' όλα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουν το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. γνωμοδότηση για οικογενειακής οικογενειακές στην Ευρώπη. Συντάκτη γνωμοδότησης η κυρία Αγιούτο. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μπορούμε να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα, η τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Non. 35. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υ... Όχι, συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 37. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ξαναρχίζει η ψηφοφορία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 46 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 η... χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Adopté. 57. Εγκρίνεται λοιπόν και περνούμε στην 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται λέει πρόεδρος. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Ε, όχι, 4 λέει η πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 χωρίς τη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Έχω την εντύπωση ότι απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 23. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχω την εντύπωση λέει η πρόεδρος ας κάνουμε όμως ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία Ψηφίζουμε την 26. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση στο σύνολό της. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 21 προς 3 και 3 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας και συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Uh,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 προφορική τροπολογία που κατέθεσε η συγγήτρια. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31. Υπέρ, Την 32 την ψηφίσαμε. Τώρα ψηφίσουμε 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λεβοτεκλό. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 με προφορική τροπολογία που κατέθεσε η συγγετρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Ε, ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση διότι δεν είναι σαφή τα αποτελέσματα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Υπέρ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 Όχι, όχι, όχι. Ναι, 48, 48. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Συγγνώμη λέει πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 47. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. 48. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55. Υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται νομίζω, αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονική επελήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μήπως μπορούν να ψηφίσουμε ο μπλοκ από την 67 έως και την 2 Όχι Άρα ψηφίζουμε χωριστά την καθεμία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73. Υπέρ Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας αν δεν έχετε αντιρρήσεις υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επελήθευση της 7 αρχίζει η ψηφοφορία Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δέκα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται Έντεκα υπέρ, κατά, αποχή. Εγκρίνεται υπέρ, κατά, αποχή εγκρίνεται 13 υπέρ κατά Εποχές. εγκρίνεται αλλά κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση της 13 υπέρ ε, συγγνώμη αρχίζει ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται 14 κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 με χωριστή ψηφοφορία ψηφίζουμε το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουν το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται θα ψηφίσουμε τώρα όλο το σχέδιο γνωμοδότησης έτσι όπως το τροποποίησαμε και ψηφίσαμε τις τροπολογίες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 21 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Χιμένεθ. Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στην ψηφοφορία. Και τώρα θα κάνουμε διάλειμμα, συνάδελφοι. Ah, we still have one vote. On a autre vote encore, c'est fini, non? Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Α, τα ψηφι... ψηφίσαμε όλες τις εκθέσεις για το gender mainstreaming προηγουμένως και μετά τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τώρα την εκθεσή του έμπολα. Ψηφίσαμε όλες τις εκθέσεις. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα στις 11. Στις 11 ακριβώς παρακαλώ αρχίζει η ακρόαση. Για τις γυναίκες οικιακές βοηθούς. Α, τούτα Θα σας δώσω μισή ώρα λοιπόν. Σα Είναι 11 η ώρα και παρεκκλήθη να αρχίσουμε αμέσως την ε, ε, συνεδρίαση. Σας παρακαλώ λοιπόν, έχετε την καλοσύνη να καθίσετε. Και καλώς ήρθατε όλες και όλοι. Θα διευθύνω τη συζήτηση. Ε, είναι και πέμπτη βέβαια πολλές και πολλοί από εσά επιθυμείτε να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Είμαι η Μέρι Χάνιμπολ από το Λονδίνο, μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών για πολλά χρόνια και με μεγάλη χαρά να λαμβάνω την διεύθυνση της συζητήσεως. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Οι ε, γυναίκες οικιακές βοηθοί και πρόσωπα που φροντίζουν εξαρτημένα άτομα πάντοτε μας απασχολούν πάρα πολύ. Είμαι βεβαίω ότι η σημερινή συνεδρίαση θα μας προσφέρει περισσότερες ιδέες αλλά και θα μας δείξει τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο των προσώπων αυτών. Έχουμε ορισμένους διακεκριμένους ομιλητές που είναι και ειδικοί στον τομέα τους. Θα ήθελα πρώτα λοιπόν να τους συστήσω έναν προς έναν ή μία προς μία. Έχετε και το πρόγραμμα, άρα γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται. Και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στο τέλος της παρουσίασης που θα κάνουν. Ο πρώτος θα είναι ο Χόρχε Καμπρίτα, από την Πορτογαλία, ερευνητής και ασχολείται με θέματα κοινωνικού διαλόγου και είναι υπεύθυνο για διάφορες ε, δραστηριότητες που έχουν σχέση και με τα ευρωπαϊκά παρατηρητήρια και, το, και την ευρωπαϊκή επιθεώρηση συνθήκων εργασίας και τώρα ασχολείται με βιομηχανικές σχέσεις και εργασία σε ε, δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες κλπ. και ζητήματα ισότητας φύλων στα πλαίσια των κοινωνικών εταίρων. Ο Χόργε έχει ήδη εργαστεί, πώς θα, το, προ... πώς θα το προφέρω τώρα το Ινστιτούτο αυτό, πάντως ένα Ινστιτούτο το οποίο έχει την έδρα του στη Λισαβόνα, η CIS, και μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων συμμετέχει και στην εθνική τους ομάδα ανταποκριτών για την οργάνωσή του αυτή. Έχει και πτυχίο ε, κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων από το Πολυτεχνείο της Λισαβόνας. Έχετε λοιπόν το λόγο εσείς ε, τώρα κύριε Καμπρίτα στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω για λογαριασμό του οργανισμού μου, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βελτίωσης των Συνθήκων Εργασίας, που με έχετε προσκαλέσει και μπορώ να εξηγήσω ορισμένα από τα συμπεράσματα των ερευνών μας ε, για τον χώρο της φροντίδας. Έχω και ορισμένες διαφάνειες. Βέβαια η οθόνη σας είναι κάπως μικρή και ίσως να μην βλέπετε καθαρά όλες τις λεπτομέρειες των διαφανειών, αλλά θα σας δώσουμε το κείμενο της ε, παρουσίασης μετά. Ελπίζω θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την ομιλία μου. Η ομιλία μου βασίζεται κυρίως σε δεδομένα από τις έρευνές μας και ιδίως από την επιθεώρηση ε, συνθήκων εργασίας Ιδίως για τις ε, οικιακές βοηθούς. Άλλες παρουσιάσεις αναφέρονται επίσης στην οικιακή εργασία. Έχουμε και σχετικές έρευνες βέβαια και εμείς. Αλλά εμείς προτιμούμε να, εγώ δηλαδή, ε, προτιμώ να περιοριστώ ε, τα πρόσωπα εκείνα που προσφέρουν φροντίδα σε εξαρτώμενα άτομα. Αυτό με ενδιαφέρει εν προκειμένου Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι ιδέες ενδεχόμενα να ληφθούν υπόψη και στις πολιτικές σας συζητήσεις. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι να δούμε την, το χάσμα που υπάρχει. Έχουμε κάνει πολλές μελέτες για τα θέματα της ισότητας των φύλων. Έχουμε κάνει και δευτερεύουσες αναλύσεις για τις γυναίκες και τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας τις οποίες αναφέρουν. Ένα Μία από τις φράσεις που ακούμε είναι ότι οι γυναίκες και άντρες απασχολούνται σε διαφορετικές θέσεις στον κλάδο, έχουν διαφορετικές συμβάσεις εργασίας, διαφορετική αμοιβή και διαφορετικούς χρόνους εργασίας. Και αυτό βέβαια ισχύει και για την προσφορά των υπηρεσιών αυτών. Κυρίως βέβαια πρόκειται για γυναίκες. Εκεί 81% εκεί απασχολούνται γυναίκες. Οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές σε δουλειές χαμηλών προσόντων. Πολύ λίγοι άντρες λοιπόν στον τομέα αυτό και οι περισσότεροι από τους άντρες αυτούς είναι μάνατζερ. Έχουν δηλαδή υψηλά προσόντα. Είναι λοιπόν πολύ έντονη η διαφορά και είναι και αντιπροσωπευτική και άλλων τομέων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Πάντως, να δούμε και τα ωράρια εργασίας ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά στοιχεία που βλέπουμε. Στον τομέα αυτό οι γυναίκες και άνδρες δουλεύουν λιγότερες ώρες. Κοιτάξτε εκεί τις ε, μπλε αυτές γραμμές που δείχνουν ιδίω ότι οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερες ώρες από το μέσο όρο σε άλλους κλάδους. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων αυτών δουλεύουν part-time, δουλεύουν σε μερικό, μερικό χρόνο εργασίας. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που βλέπει κανείς. Αν δούμε τώρα τις προτιμήσεις ωραρίου εργασίας, θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες προτιμούν μάλλον να δουλεύουν λιγότερες ώρες, ακόμα λιγότερες από ό,τι ήδη δουλεύουν, ενώ οι άντρες προτιμούν να δουλεύουν περισσότερες ώρες. Δεν έχουμε καμία εξήγηση γι' αυτό, ίσως μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανές εξηγήσεις και με τους άλλους ειδικού εδώ, αλλά είναι μια έντονη διαφορά που φαίνεται και στο πίνακα που δείχνω και υποθέτουμε ότι αυτό εφαρμόζεται και στις οικιακές βοηθούς. Αυτό ισχύει δηλαδή και για τις οικιακές βοηθούς. πάλι στον τομέα του, των ωραρίων εργασίας. Οι άνθρωποι στον κλάδο που συζητούμε δουλεύουν λιγότερο, σε λιγότερο τυπικά ωράρια και λιγότερο τακτικά ωράρια. Όταν λέω τυπικά ωράρια, μιλώ για καταστάσεις όπου οι άνθρωποι δουλεύουν και Σάββατα, Κυριακές, βράδια και νύχτες. Και αυτό ισχύει και για άντρες και για γυναίκες, βέβαια. Δεν υπάρχει επομένως Ε, μιλούμε για ανθρώπους που, δουλεύουν τις ίδιες ώρες κάθε μέρα, τις ίδιες μέρες κάθε εβδομάδα, με ωράρια καθορισμένα για έναρξη και τέλος της εργασίας. Και αυτό ισχύει και για τους άντρες ξανά και για τις γυναίκες. Και πάντα σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Πάλι τώρα η ισορροπία μεταξύ επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής. Πάλι βλέπετε εδώ ότι οι γυναίκες που δουλεύουν στον κλάδο αυτό έχουν λιγότερο καλή ισορροπία μεταξύ δηλαδή εργασιακών υποχρώσεων και κοινωνικών οικογενειακών υποχρώσεων. Είναι λιγότερο καλή από το μέσο όρο σε σχέση με τους άλλους κλάδους. Και αν δείτε και την γαλάζια στήλη που είναι για τους άνδρες, θα δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι η σχέση μεταξύ του αυτόνομου χαρακτήρα και της εντατικότητας της εργασίας. Ανάλυση που μπορούμε να την κάνουμε βασισμένη στα δεδομένα της επιθεώρησης των συνθήκων εργασίας, γιατί η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών δείχνει και πού βρίσκεται το στρες του εργαζόμενου. Εάν κάποιος δηλαδή δουλεύει σε κάποιο βαθμό εντατικότητας χωρίς να έχει έλεγχο για τη δουλειά που κάνει, τότε αντιμετωπίζει συχνότερα και περισσότερα προβλήματα από το στρες. Θα δείτε εδώ ότι και άνδρες και γυναίκες στη διαφάνεια αυτή, βλέπετε βέβαια και άλλα πράγματα που σχετίζονται με την ηλικία, με το μέγεθος του χώρου εργασίας, αλλά θα δείτε εκεί άνδρες και γυναίκες ότι βρίσκονται κάτω αριστερά, στο κάτω αριστερό τρίτο. Και θα δείτε επίσης ότι αυτό αναφέρεται σε έναν τύπο εργασιών που λέγονται παθητικές εργασίες. Πρόκειται δηλαδή, επειδή πρόκειται για δουλειές που δεν αποτελούν πρόκληση, έχουν μια απογοήτευση, μια ε, απογοήτευση από τη δουλειά και αυτό είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του τομέα αυτού σε σύγκριση με άλλους. Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των ε, συνθήκων εργασίας είναι και το κοινωνικό περιβάλλον. Το κοινωνικό περιβάλλον εδώ για μας σημαίνει ότι έχει σχέση με την κοινωνική υποστήριξη που δίνουν οι άλλοι συνάδελφοι, που δίνουν οι προϊστάμενοι και μια γενική αίσθηση των ανθρώπων, αν δηλαδή αισθάνονται ότι υποστηρίζονται αρκετά μέσα στη δουλειά που κάνουν ή όχι. Πάλι ο τομέας αυτός δείχνει ότι είναι πολύ περιορισμένη η υποστήριξη αυτή από το κοινωνικό περιβάλλον σε σύγκριση με άλλους κλάδους. Και αυτό λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ε, κλάδου αυτού. Άλλο θέμα ανισχυτικό για τον ε, κλάδο αυτό είναι και η έκθεση σε φυσικούς κινδύνους. Με τα δεδομένα που έχουμε μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε τριών ειδών ε, φυσικούς κινδύνους. Για παράδειγμα αν χρειάζεται κανείς να σηκώνει ε, μεγάλα βάρη, ένα ε, βαρύ άνθρωπο για παράδειγμα να τον σηκώσει κτλ. Επίσης η επαφή με χημικά, χημικές ουσίες ή φάρμακα κλπ. Και επίσης οι συνθήκες του περιβάλλοντος, θόρυβος, θερμοκρασία κλπ. Αυτό το τελευταίο δεν δείχνει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το μεσονόρο. Υπάρχει ωστόσο ένα μια χαρακτηριστική διαφορά, διότι η έκθεση σε κινδύνους από κίνηση ή από χημικά φάρμακα κτλ. είναι πολύ ψηλότερη από τον μέσον όρο. Και αυτό εδώ είναι ένα σημείο ανησυχίας, ιδίω για γυναίκες και ιδίω για γυναίκες σε χειρονακτικές εργασίες, εργασίες δηλαδή λιγότερο εξειδικευμένες εργασίες, που απαιτούν λιγότερα προσόντα. Με απλά λόγια δηλαδή, αν δείτε και την διαφάνεια, θα δείτε ότι οι γραμμές αυτές είναι πολύ υψηλότερες για τις γυναίκες. Βλέπετε λοιπόν ότι για τον κλάδο αυτό και ιδίω για τις γυναίκες σε χειρονακτικές απασχολήσεις ο, κίνδυνος αυτός είναι πολύ υψηλότερος και για κινδύνους δηλαδή βιο, βιολογικούς και χημικούς και για κινδύνους από κίνηση όπως για τη μεταφορά βαριών φορτίων. Άλλο θέμα είναι η απουσία το absenteeism είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσον όρο. Προσπαθήσαμε αυτό να το κατανοήσουμε καλύτερα. Όταν κάνουμε έλεγχο για ισότητα μεταξύ φύλων, ηλικίες κλπ. Εκεί βέβαια θίγονται κυρίως γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Άλλο είναι το θέμα των προβλημάτων υγείας. Ζητούμε από τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους να αναφέρουν αν έχουν προβλήματα υγείας και έχουν και ένα κατάλογο. Αν πάρετε τον αριθμό των προβλημάτων υγείας, βλέπετε κατά μέσον όρο οι άνθρωποι εκεί να αναφέρουν περισσότερα προβλήματα υγείας σε σύγκριση πάντα με το μέσον όρο, που δεν σχετίζονται βέβαια πάντα άμεσα με την εργασία τους, αλλά πάντως οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι αναφέρουν περισσότερες ασθένειες. Συνοπτικά λοιπόν βλέπουμε ότι κυρίως εκεί απασχολούνται γυναίκες στον τομέα φροντίδας, ε, δηλαδή εξαρτώμενων προσώπων κλπ. Είναι μη τυπική εργασία, είναι χαμηλή η ένταση εργασίας και είναι μάλλον παθητικού τύπου εργασίες που οδηγούν βέβαια σε μια απογοήτευση των ανθρώπων που, που δουλεύουν στη, στον τομέα αυτό. Είναι χαμηλό επίπεδο το κοινωνικό περιβάλλον, υψηλό Υψηλό ωστόσο το επίπεδο έκθεσης σε κινδύνους βιολογικούς, χημικούς κλπ. Και τέλος υψηλό το επίπεδο των απουσιών και επίσης υψηλό το επίπεδο των ασθενειών ή άλλων προβλημάτων υγείας που αναφέρουν οι εργαζόμενες. Σε αυτή τη διαφάνεια θα, πολύ, πω πολύ γρήγορα γιατί είναι από μια έκθεση που είχαμε συντάξει το 2006 με έρευνα για την απασχόληση στον κοινωνικό τομέα στην Ευρώπη. Ήδη τότε είχαμε δει ότι πρόκειται για τομέα χαμηλού κύρους, πάλι εκεί κυρίως γυναίκες, χαμηλή ορατότητα που θεωρείται ότι είναι κάτι για ανθρώπους με, χαμηλό, με χαμηλά προσόντα, είναι part-time και ούτω καθεξής. Η κατάσταση λοιπόν εξακολουθεί να είναι ίδια από τότε, σχεδόν 10 χρόνια μετά, το 2006 είμαστε τώρα 2015. Έχουμε πάντα σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ελπίζω λοιπόν ότι σας έδωσα κάποιες ε, πρόσθετες πληροφορίες και κάποιες πτυχές όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα των εργασιών αυτών. Και κυρίως ότι αν είναι δυνατόν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Ίσως έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, αλλά οδηγούμε πλέον στο τελικό συμπέρασμα. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι για να αντιμετωπιστεί αυτός ο διαχωρισμός των φύλων στον τομέα αυτό θα πρέπει να δούμε αυτή την υποβάθμιση της ε, εργασίας των γυναικών και αυτά τα στερεότυπα που οδηγούν κορίτσια και αγόρια σε ένα συγκεκριμένο είδος εργασίας. Βέβαια αυτό ισχύει και σε άλλους κλάδους, αλλά σίγουρα ισχύει εδώ, έχει σχέση με την εκπαίδευση που έχει ο καθένας και με τον τρόπο αυτό οδηγείται στο να επιλέξει το, την εργασία του. Υπάρχουν και τα άτακτα ωράρια εργασίας που ίσως έχουν πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην, στην υγεία των εργαζόμενων. Και αυτό παίζει λοιπόν ένα σημαντικό ρόλο, ιδίως για τις γυναίκες στον κλάδο. Μέτρα τώρα για την βελτίωση της ποιότητας της εργασίας. Αν πάρουμε αυτά που έχουν, όπως είπα προηγουμένως, αρνητικό χαρακτήρα και αν θέλουμε να τα βελτιώσουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι βελτιώσεις αυτές να ισχύσουν και για γυναίκες και για άντρες. Και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας απασχόλησης χαμηλού επίπεδου για αυτούς που πρωτομπαίνουν στο επάγγελμα. Πρέπει να βρεθούν τρόποι που τονώνουν και βελτιώνουν την ποιότητα της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας και τέλος δύο λόγια για την βελτίωση της διαχείρισης και της οργάνωσης της εργασίας. Υπάρχουν τρόποι εκεί εξυγχρονισμού για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο αυτό. Υπάρχουν και σχετικές δημοσιεύσεις, τις βλέπετε σε αυτή τη ε, διαφάνεια και μάλιστα ορισμένες από τις δημοσιεύσεις αυτές τις έχω βάλει στο τραπέζι εκεί κοντά στην έξοδο. Αυτές θα πω και σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ πληρέστατη παρουσίαση. Θίξατε πολλά θέματα. Πριν προχωρήσουμε στους επόμενους φιλοξενούμενους μα θα πάρουν το λόγο, να ζητήσω από την εισηγήτρια την κυρία Κούνεβα να πει μερικά λόγια για το θέμα εν γέννη, αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε από το κοινό το θέμα το προσωπικό οικιακής εργασίας. Η οικιακή εργασία αποτελεί ένα φαινόμενο με πολλές διαστάσεις. Συνδέεται με ζητήματα που σχετίζονται με μεγάλο βαθμό με την εθνικότητα, την ηλικία και το φύλλο των εργαζομένων. Η συντριπτική πλειοψηφία του εργαζομένου πληθυσμού στα σπίτια αποτελείται από γυναίκες, μετανάστριες, ορισμένες με τις οποίες είναι μέση ηλικία και πάνω. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, 53 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω εργάζονται σταθερά και συστηματικά στο πλαίσιο ενός νοικοκυριού ενός σπιτιού το 83% αυτών των εργαζομένων είναι γυναίκες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η διάσταση του φύλου για το φαινόμενο της οικιακής εργασίας και αυτό είναι τόσο σημαντική που η έκθεση θα συνταχθεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης και Οικονομικών Θεμάτων. Τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια της κρίσης που αποδόμησε το κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές παροχές η έξοδος στη νόμιμη αγορά εργασίας έγινε πιο δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις ήταν απαγορευτική για μια γυναίκα. Η κατάσταση αυτή ανάγκαζε πολύ κόσμο, κυρίως γυναίκες, να στραφούν σε άπειτες μορφές εργασιακών σχέσεων σε οικιακά περιβάλλοντα που όμως λόγω της φύσης τους δύσκολα οριοθετούνται. Η οικιακή εργασία ακριβώ λόγω της ιδιόμορφης και συνήθω μη ρυθμισμένης φύσης της οδηγεί σε πολύπλευρο αποκλεισμό. Αποκλεισμό από το σύστημα πρόνοιας από τη φροντίδα των ίδιων των εργαζομένων των παιδιών τους από τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα από την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Οι γυναίκες που εργάζονται σε οικιακό περιβάλλον επειδή δεν έχουν χαρτιά ή δεν μπορούν να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά την ε, εργασία τους επιδιώκουν συχνά σε ένα αόρατο συχνά να είναι αόρτες προκειμένου να επιβιώσουν. Στις χώρες του Νότου οι μετανάστες καλύπτουν αυτό που αποτελείται χάσμα υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών ισότητας των φύλων. Οι πολιτικές αυτές που θα βοηθήσουν την έξοδο των γυναικών στην αγορά εργασία, η φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, άτομα με αναπηρία δεν εφαρμόζονται κυρίως σε αυτές τις χώρες και το κενό το καλύπτουν οι μετανάστες εργαζόμενες στο σπίτι που αναλαμβάνουν την φροντίδα μέων της οικογένειας των γυναικών που θέλουν να δουλέψουν. Πρόσφατα συνέβη στην Ελλάδα ένα ακόμη φρικιαστικό περιστατικό κακοποίησης μιας οικιακής εργαζόμενης από τη Βουλγαρία, της Αναστασίας η οποία φρόντιζε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Κατηγορώντας την Αναστασία πώ έκρυψε χρήματα, ο ιό τη και οι δύο φίλοι του την ξυλοκόπησαν, την βασάνιζαν και την εγκατάλειψαν αιμόφερτη σε, ερεμικό, σε ειρημική περιοχή. Για να μην νιώσει ξανά ανα, ανεπεράσπιστη και αόρατη Αναστασία για να πάψουν να είναι αόρατοι για το κράτος και τις υπηρεσίες εργαζόμενοι στο σπίτι αλλά και να αποτρέψουμε εργοδότες οικιακών βοητών να μεταμορφώνονται σε σκληρούς και, ανα... και απάνθρωπους αφέντες είναι ανάγκη να εργαστούμε από κοινού ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές που τα προστατεύουν τους εργαζόμενους ώστε να είναι ασφαλείς και να εξασφαλίζουν τα ατομικά και συλλογικά τους δικαιώματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Oh, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στους φιλοξενούμενους μας και επόμενος είναι ο κύριος Ιορδάνης Ψημένος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα και είναι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο των Αθηνών από το 2006 και υπήρξε και ελέκτορας της κοινωνιολογίας εκεί και διδάσκει βιομηχανική κοινωνιολογία και συγκριτική κοινωνιολογική πολιτική και την κοινωνιολογία της μετανάστευσης. Εστιάζεται το έργο του κυρίου σε θέματα της συμμετοχής των εργαζομένων ε, στη μεταναστευτικό αποκλεισμό και έχει συγγράψει διάφορα έγγραφα όπως η παγκοσμιοποίηση και η συμμετοχή των εργαζομένων η μετανάστευση τα Βαλκάνια, η μετανάστευση εκκλησία στην Ευρώπη, η μετανάστευση εργαζόμενη, κοινωνική προστασία, η περίπτωση των γυναικών από την Ουκρανία και την Αλβανία. Δημοσίευσε πολλά άρθρα όσον αφορά τον αποκλεισμό των Ουκρανών, των Πολωνών και των Αλβανών εργαζομένων ε, και εργαζομένων στις κατασκευαστικές στις κατασκευές, ε, ανισότητες ε, και διάφορα θέματα του 2013. Επίσης είναι μέλος αρκετών επιστημονικών επιτροπών και έχει κάνει εξολογήσεις για διάφορα ειδικά επιστημονικά περιοδικά. Επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνιολογίας και της Διεθνούς Ενώσεως Κοινωνιολογίας και, έγραψε διάφορα μοναγράφα για κοινωνικές ανισότητες στην σύγχρονη Ελλάδα. Και πρόκειται να μας μιλήσει για τις γυναίκες μετανάστριες ε, τις εργαζόμενες και για το πώς επηρεάζεται, ε, επηρεάζονται οι σχέσεις τους, η οικογενειακή του ζωή και από το περιβάλλον αυτό. Ευχαριστώ λέει ο που με καλέσατε να μιλήσω σε αυτό το πάνελ. Θα μιλήσω ελληνικά ούτως ώστε να διευκολυνθούμε όλοι. Α, Υπάρχουν 52,6 εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο και άντρες που δουλεύουν ως οικιακές και οικιακοί βοηθοί, οικιακές εργάτριες, οικιακοί βοηθοί και ε, ε, πιστεύω ότι ε, όλα τα ντοκουμέντα δείχνουν ότι έχουμε δύο βασικές ιστορίες να πούμε οι οποίες ίσως βοηθήσουν περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει τις κατάλληλες πολιτικές. η μία ιστορία είναι η γυναικεία εργασία στο σπίτι και το πώς η μετανάστευση και η οικιακή, η εργασία ουσιαστικά εμποδίζουν την κοινωνική κινητικότητα των οικιακών εργατριών. Σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι εργάτριες είναι τεράστια. Η εκμετάλλευση τεράστια και μέσα σε αυτά τα στοιχεία που έχω δώσει στο, στην ομιλία μου και πιστεύω ότι ε, σύντομα θα έχετε στη διάθεσή σας θα καταλάβετε ότι μιλάμε για απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Μέσα όμως σε αυτές τις 52,6 εκατομμύρια ιστορίες γυναικών και ανδρών που δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί ή οικιακοί εργάτες και εργάτριες υπάρχει μια ιστορία που κατά τη γνώμη μου από το 1991 έως σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχνά να πει. Ποια είναι αυτή η ιστορία, είναι η ευρωπαϊκή διάσταση της οικιακής εργασίας των μεταναστριών. Α, υπάρχουν τρία βασικά θέματα τα οποία ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κάθε χώρα ξεχωριστά ξεχνά να μελετήσει. Το πρώτο είναι η ιστορική διάσταση της μετανάστευσης και της οικιακής εργασίας στην Ευρώπη. Ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα για το οποίο ίσως θα πρέπει επιτέλους μετά από 25 χρόνια παραμονής των γυναικών στο ευρωπαϊκό έδαφος ως οικιακές εργάτριες θα πρέπει να υποθεί. Το δεύτερο θέμα το οποίο επίσης μας αφορά έχει να κάνει ε, ε, ε, αξιότιμα μέλη της Ευρωβουλής έχει να κάνει με την οικονομική και κοινωνική πολιτική των ευρωπαϊκών μελών των κρατών οι οποίες φαίνεται, αυτή η πολιτική φαίνεται να διαμορφώνει όχι καλές συνθήκες για την εξέλιξη των ανθρώπων αυτών. Στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου σύμφωνα με υπολογισμούς 4 εκατομμύρια ε, νόμιμοι, νόμιμες μετανάστες οικιακές εργάτριες αν συνυπολογίσουμε και από διάφορα, ε, διάφορες εκθέσεις το πόσες γυναίκες είναι χωρίς χαρτιά και δεν καταγράφονται από καμία κοινωνική ή στατιστική υπηρεσία ε, πιστεύω ότι ο αριθμός ξεπερνά σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών τα 7,7 εκατομμύρια. Το τρίτο θέμα το οποίο επίσης μας αφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση είναι οι πολιτικές που αφορούν την, την πρόνοια, την προστασία, την κοινωνική κινητικότητα και την οικογενειακή επανένωση. Θα σταθώ, αν μου επιτρέπετε, σε αυτά πολύ σύντομα γιατί ξέρω ότι έχω μόνο 8 λεπτά και ελπίζω να τα καταφέρω. Ένα βασικό θέμα το οποίο φαίνεται από τις μελέτες μας που έχουμε διεξάγει από το 1991 μέχρι και σήμερα είναι ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που δημιουργεί την οικιακή εργασία σε πρώτο επίπεδο και εγκλωβίζει την οικιακή εργάτρια στο περιθώριο της κοινωνικής προστασίας είναι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις. Δυστυχώς θα δείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργατριών ισχωρούν στην οικιακή εργασία και εγκλωβίζονται σε αυτή λόγω της αδυναμίας τους να επιβιώσει η οικογένειά τους. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε περισσότερες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δυστυχώς συνδέονται με την νομιμοποίηση των μεταναστών και με την εργασία. Και τα δύο δυστυχώς διαμορφώνουν ένα κοινωνικό φράγμα απέναντι στην δυνατότητα μιας γυναίκας μετανάστριας να ψάξει αλλού δουλειά. Το δεύτερο το οποίο φαίνεται από τις μελέτες τις οποίες έχουμε διεξάγει εδώ και 25 χρόνια στη χώρα μας αλλά και διεθνώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι μετά από 10 χρόνια παραμονής στην οικιακή εργασία πολλές από τις μετανάστριες φαίνεται να αδυνατούν ή και να μην μπορούν πλέον οικειοθελώς να συνδεθούν με την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό εξηγείται και αν μου δώσετε αργότερα την δυνατότητα θα προσπαθήσω με το διάγραμμα το οποίο έχω εδώ να σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Ε, το τρίτο θέμα για την κοινωνική πρόνοια αφορά την ε, δεκαετία περίπου 2009 μέχρι σήμερα όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο ανάπτυξης ξανά μιας εργοδοτικής ασφάλισης εντός της οικιακής εργασίας και εντός της οικογένειας με άτυπες μορφές. Θα προχωρήσω με το θέμα της κοινωνικής κινητικότητας και ειδικότερα της καριέρας. Επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κάθε χώρα ξεχωριστά ανακαλύπτουμε συνεχώς σε όλες μας τις μελέτες, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλοι συνάδελφοι, ότι μια βασική παράμετρος εισόδου των, των μεταναστριών γυναικών εισόδου στην οικιακή εργασία είναι η αδυναμία τους να αναγνωρίσουν βασικά εκπαιδευτικά και άλλα εργασιακά, ε, άλλες εργασιακές δεξιότητες. Το γιατί συμβαίνει αυτό σε κάθε χώρα ξεχωριστά και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αν υπάρχει χρόνος αργότερα. Όμως δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας που ουσιαστικά διαμορφώνει την οικιακή εργασία. Φαίνεται ο δημόσιος τομέας, ο κρατικός τομέας να είναι εκείνος που διαμορφώνει ενεργατικό δυναμικό χωρίς προσόντα. Οι περισσότερες από τις γυναίκες που εμείς τουλάχιστον από το 1991 μέχρι σήμερα έχουμε πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις όχι μόνο είναι αυτό που λέμε με αυξημένες δεξιότητες αλλά θα μπορούσαν ως ανθρώπινο κεφάλαιο να προσφέρουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταυτού δυστυχώς βρίσκονται στην οικιακή εργασία και φροντίδα. Το δεύτερο όσον αφορά με την κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα και την καριέρα, το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουμε ουσιαστικά ένα μεγάλο πρόβλημα με τα θέματα της μετεκπαίδευσης των γυναικών. Τα περισσότερα προγράμματα δεν επιτρέπουν την είσοδο σε αυτά τα προγράμματα λόγω ακριβώς και της βίζας, της έλλειψης βίζας αλλά λόγω και της αδυναμίας των γυναικών να αποκοπούν από το επάγγελμά τους για οικονομικούς λόγους. Πάω κατευθείαν στο τελευταίο θέμα το οποίο αφορά την οικογενειακή σχέση και τις οικογενειακές σχέσεις των γυναικών. Ε, εδώ διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των γυναικών αποκόπτεται και από την οικογένειά του αλλά και συνδέεται με τις οικογένειες της, ε, ε, της, του ιδιωτικού νοικοκυριού. Αυτό τι σημαίνει σημαίνει ακριβώς ότι έχουμε ένα τεράστιο δέσιμο των γυναικών αυτών και σε οικονομικό αλλά και σε φιλικό επίπεδο μόνο με την εργοδοτική οικογένεια και που κατ' επέκταση διαμορφώνει ένα πλαίσιο ανυπαρξίας ή μη δυνατότητας του κράτους να παρέμβει στην κοινωνική προστασία και εξέλιξη των γυναικών στις χώρες εισόδου. Ε, τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι η κρίση σήμερα στην Ελλάδα μας δείχνει ότι πολλές οικογένειες αναγκάζονται και μένουν μόνες τους, δηλαδή γυναίκες με παιδιά στην Ευρώπη, ενώ οι άνδρες τους μεταναστεύουν για αναζήτηση μιας καλύτερης εργασίας. Αυτό βεβαίως δημιουργεί στην Ευρώπη νέα προβλήματα μονογονεϊκών οικογενειών με ίσως απροσδόκητες κοινωνικές καταστάσεις και εκρήξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ήμουν μέσα στο πλαίσιο του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έθιξε πολλά σημεία. Η επόμενη ομιλήτρια θα μας μιλήσει για το Διεθνή Οργανισμό Αργασία για την σύμβαση των οικιακών εργατών και την προστασία των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κυρία Κλέρ Κουρτέι που είναι η διευθύντρια του, της αντιπροσωπείας του οργανισμού στις Βρυξέλλες και εργάστηκε στην Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, στον ΟΗΕ, στον ΟΣΕ και στην Κολομβία και θα μας ξαναμιλήσει για 8 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σα. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Η σύμβαση 189 του Διεθνού Γραφείου Εργασία για τι Οικιακέ Βοηθού εγκρίθηκε με την συνδρομή όλων των οργανώσεων των σχετικών. Ο κύριος στόχος σύμβαση είναι να παράσχει προστασία και δικαιώματα στους οικιακές βοηθούς που είναι μία από τις κατηγορίες εργαζομένων με την μικρότερη προστασία που υπάρχει στην Ευρώπη και εκτός. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ορίζεται ως οικιακή βοηθός το άτομο το οποίο κάνει οικιακές εργασίες στα νοικοκυριά που ασχολείται με την βοήθεια στο σπίτι και είναι σημαντικό να πούμε ότι στην πράξη η διαχωριστική γραμμή μεταξύ άτομου που φροντίζει κάποιο άλλο εξαρτώμενο άτομο και εκεί βαθμού είναι αρκετά ασαφής. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν διάφορα μέτρα ώστε να μπορέσει να αποσαφινιστεί η θέση αυτή. Η συμφάνιση λέγει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες όσον αφορά την αμοιβή, κοινωνική προστασία, ασφάλεια στο σπίτι και τις ώρες εργασίας που πρέπει να συμβαδίζουν με τους κανόνες που ισχύουν για την εκάστοτε χώρα για όλους τους εργαζόμενους. Επίσης προστατεύεται το δικαίωμα των εργαζομένων αυτών να αποτελέσουν μέλος ενός εργατικού συνδικάτη. Όσον αφορά την οπτική γωνία του ε, δύο φίλων. Πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των κοινωνικών βοηθών που είναι κυρίως γυναίκες και όλων των άλλων εργαζομένων που προστατεύει ο νόμος. Έτσι δίδεται μια ιδιαίτερη αξία σε αυτούς τους και σε αυτές τις εργαζόμενους και καθορίζει ότι η αμοιβή τους, η αμοιβή τους θα πρέπει να είναι ίση με οποιοδήποτε άλλο εργαζομένο. Σύμφωνα με τις έρευνες που έγινε το 2010 υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2,5 εκατομμύρια τέτοιου είδου οικιακοί εργαζόμενοι βάσει του ορισμού που δίδεται από το δύο οργανισμό εργασία και σύμφωνα με εθνικέ στατιστικέ μα παράγουν τα κάτι μέλη. Δεδομένου όμω ότι υπάρχουν ε, άτυπε τέτοιου είδου μορφέ εργασία και δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, θα πρέπει να σε οι Περισσότεροι οικιακοί βαθμοί ε, υπάρχουν σε απόλυτου αριθμού ε, τέτοιοι εργαζόμενοι στην Ισπανία, 750.000, 600.000 στην Ιταλία και κάποιες λιγότερες εκατοντάδες τέτοιες εργαζόμενες στην εργασία. Μιλώ για οικιακές εργαζόμενες ε, γυναίκες. Από αυτές τις 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενες, το 2.200.000 είναι γυναίκε, το 80%. Πρόκειται λοιπόν για ένα τομέα στον οποίο κυρίω εργάζονται γυναίκε. Και η ιδιαιτερότητα αυτή τη εργασία είναι όχι ότι κυριαρχείται από γυναίκε, αλλά κυρίω και από εργοδότριε γυναίκε. Πράγμα το οποίο είναι παραδοσιακό του ρόλου της γυναίκας και του άντρα στα ευρωπαϊκά ε, νοικοκυριά. Και οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται στην χώρα εργασία είναι επίσης υπεύθυνε για τις γυναίκες οι οποίες θα αναθέσουν τον οικογενειό. Ε, τώρα, ποιο είναι το επίπεδο επικύρωσης της σύμβασης αυτής στην Ευρώπη. Ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχουν τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ε, επικυρώσει την ε, ε σύμβαση καθώς και η Ελβετία και το Βέλγιο είναι πολύ κοντά στην τελικό στάδιο τη επικαιρία. Θα σα εξηγήσω γιατί είναι πόσο σημαντικό για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε να επικαιρώσουν τη σύμβαση αυτή. Για δύο κυρίους λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι πρόκειται για μια κατηγορία στην οποία όλο και περισσότερου εργαζόμενου έχουμε. Εάν δούμε τα ποσοστά αυτών των ε, εργαζομένων ε, σε σχέση με την απασχόληση στην Ευρώπη, θα δούμε ότι οι περισσότερες, όπως σας είπα, που έχουν τέτοιου είδους εργαζόμενες είναι η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, αλλά για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουμε ποσοστό της τάξης του 1% περίπου. Όμως πρέπει να σας πω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ποσοστά αυτό από το 1995 μέχρι το 2010. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα στην οποία ο αριθμός των οικιακών εργαζομένων μειώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά σύμφωνα με κάποιες έρευνες που έγιναν, αυτό ίσως έχει σχέση με το γεγονός ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οικογένειες όλο και περισσότερο ε, προσφεύγουν σε, στις ε, νέες κοπέλες ΟΠΕΡ ως εναλλακτική λύση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο αριθμό των εργαζομένων, των οικιακών εργαζομένων, όλο και περισσότερο θα αυξάνεται και θα ήθελα να σα εξηγήσω σύντομα για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν δύο δημογραφικέ τάσει, οι οποίε ε, μας οδηγούν σε αυτή την ε, παρατήρηση. Η Γύρανση του πληθυσμού και το ότι όλο και περισσότερε γυναίκε εργάζονται στην αγορά εργασία. Οι δύο τάσεις αυτές ε, δημιουργούν όλο και περισσότερη ζήτηση για οικιακέ εργάτριες. Υπάρχει όμως τώρα μία αντίφαση όσον αφορά την απασχόληση. Αφενό, οι περισσότερε πολιτικέ στην Ευρώπη ενθαρρύνουν τι γυναίκε όλο και περισσότερο να μπουν στην αγορά εργασία και απ' την άλλη, σε εθνικό επίπεδο, οι περικοπέ στον κοινωνικό τομέα, ε, κυρίω ε, για την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, δεν καλύπτουν τι δαπάνε για τέτοιου είδου εργαζόμενου. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει κανεί ε, να προσπαθήσει από μόνος του να βρει μια, ένα άτομο που θα φροντίσει τα άτομα αυτά της οικογένειας. Ε, στις σκανδιναβικές χώρες. Δεν θεωρείται ίσως πάρα πολύ σωστό να έχει κανείς τέτοιους άτομα. Εκεί, σύμφωνα με τις δικές μας έρευνες, στην Δανία και στην Σουηδία το ποσοστό είναι κάτω από 1%. Πράγμα το οποίο έχει να κάνει με την ε, γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη από το κράτος για την φύλαξη των παιδιών και των ηλικιωμένων. Ε, Επί προσθέτως, πρέπει να πω ότι υπάρχει και το θέμα της προσφοράς. Ίσως η κατάσταση να διαφέρει από μία χώρα στην άλλη, αλλά σφαιρικά έχουμε να κάνουμε με φτηνό, ανειδίκευτο, εργατικό, δυναμικό, το οποίο είναι το μεγάλο ποσοστό των οικιακών εργατριών. Τελευταίος, λόγος για τον οποίο πρέπει να επικυρωθεί η πρόσβαση είναι για να μπορέσει να δοθεί ένα πιο επίσημο ε, καθεστώς και πιο πλαισιωμένο για τους εργαζόμενους ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Κάποιες εκτιμήσεις λέγουν ότι υπάρχει και σε ποσοστό 70 με 80% εργασία η οποία δεν συνάδει με τους κοινωνικούς ε, κανόνες και τις πολιτικές που πρέπει να ισχύουν. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν με επίσημα ίσως δηλωμένους εργαζόμενους. Συμπερασματικά, η σύμβαση αυτή, η 189, προσπαθεί να βελτιώσει τους όρους ε, απασχόλησης αυτών των εργαζομένων και θα θέλαμε να ζητήσουμε σε, από εσά να ζητήσετε από όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν την τόσο σημαντική σύμβαση αυτή του Διεθνού Οργανισμού Εργασία. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, σα ευχαριστώ και εγώ. Μα δώσατε τροφή για σκέψη. Ιδίω για το τι μπορούμε να κάνουμε για να πείσουμε τις χώρες μας να κυρώσουν την ε, σύμβαση του ILO. Τώρα η κυρία Μαρή Μπετρό από τη Γαλλία για κοινωνική καινοτομία. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οικιακών Βοηθών, μέλος του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου στη Γαλλία. Έχει μάλιστα συγγράψει διάφορα βιβλία για τα θέματα αυτά και έχει παρασημοφορηθεί κιόλα. Κυρία Λεβό, λοιπόν. Να σας τα πω στα γαλλικά, λοιπόν. Να ευχαριστήσω πρώτα τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών την Πρόεδρο και την κυρία Εισηγήτρια. Για να επανέλθω λίγο στις προηγούμενες παρεμβάσεις, να πω ότι στη Γαλλία η κατάσταση των γυναικών είναι κάπως ιδιαίτερη σε ό,τι αφορά την ε, οικιακή εργασία και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Πρώτα ορισμένα δεδομένα. τα οικιακά, συνολικά και φροντίδα των παιδιών, ανέρχονται σε 60 δισεκατομμύρια όρων μη αμοιβόμενων. Πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν το καθόριστο εθνικού προϊόντος. Δύο φορές περισσότερο οι γυναίκες εργάζονται στα οικιακά και αναλαμβάνουν και τις πιο επαναληπτικές και ρουτινιάρικες δουλειές στον τομέα αυτό. Η πρακτική εξελίσσεται και τα τελευταία 25 χρόνια βλέπουμε μια τάση σε ό,τι αφορά τον χρόνο που αφιερώνουν οι γυναίκες στα οικιακά, στις οικιακές εργασίες. Συγκριτικά, η πρόοδος, ε, συγκρίνεται μάλιστα και η πρόοδος των γυναικών στη Γαλλία στο επάγγελμα. Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γονιμότητα της Γαλλίδας γυναίκας που είναι στα δύο παιδιά περίπου ένα γυναίκα και στα 60% η συμμετοχή στο επάγγελμα. Η κατάσταση αυτή που μπορεί να θεωρηθεί και καλή πρακτική επιτρέπει να απαντήσω στα όσα άκουσα προηγουμένως για το γεγονός ότι τα οικιακά δεν υπάρχουν πλέον ως όρος στην Γαλλία. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και ένας όρος δύσκολο να χρησιμοποιηθεί σήμερα. Μιλούμε για περισσότερο για απασχολήσεις οικογενειακές και για διάφορα επαγγέλματα. Εδώ έχουμε βασιστεί σε διάφορα πράγματα, σε διάφορους μοχλούς. Αύξηση των κέντρων υποδοχής νεαρών παιδιών. Επίσης φροντίδα για τους ηλικιωμένους και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα βέβαια η εξέλιξη των ε, υγειακών επαγγελμάτων. που είναι και άξονας της κοινωνικής πολιτικής, η οποία έχει συμβάλει αφενός στην αναγνώριση των ε, φροντίδων και στην αναγνώριση των φροντίδων αυτών σαν ξεχωριστό επάγγελμα. Παραδοσιακά λοιπόν αυτά τα πράγματα θεωρούνται χωρίς αξία, αυτά είπαν και οι προηγούμενοι, ωστόσο η φροντίδα και τα οικιακά στη Γαλλία σιγά σιγά φεύγουν από την ανεπίσημη οικονομία τα τελευταία 30 χρόνια και μπαίνουν σε δηλωμένα επαγγέλματα πλέον. Πρόκειται για μια απλούστευση για την δήλωση από την οικογένεια των επαγγελμάτων αυτών. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένας άξονας ισχυρός στήριξης των ε, δραστηριοτήτων αυτών με την προϋπόθεση ότι είναι δηλωμένα και τρίτο και μία πολιτική κινήτρων προς μια κίνηση προς έναν επαγγελματισμό. Όπως είπατε και πριν, πρόκειται για γυναίκες εργοδότριες που απασχολούν γυναίκες εργαζόμενες. Αυτό παραμένει μια πραγματικότητα. έχουμε 3,6 εκατομμύρια που, ε, νοικοκυριά που απασχολούν οικιακές βοηθούς ή για την φροντίδα των παιδιών, ένα εκατομμύριο οικογένειες περίπου απασχολούν 500.000 περίπου ε, βοηθούς. Ένα εκατομμύριο πρόσωπα σήμερα στη Γαλλία έχουν φροντίδα στο σπίτι από βοηθούς και αυτά έχουν λάβει και διαφορετικά ονόματα. Η σημειολογία λοιπόν στη Γαλλία είναι διαφορετική. Η βάση του έργου μας βασίζεται και σε κάποια στοιχεία καινοτομίας, νέοι τρόποι οργάνωση της εργασίας, είτε για την εργασία εκτός του σπιτιού είτε και εντός του σπιτιού, θεωρούμε σήμερα ότι ένα σημαντικό στοιχείο της αλλαγής των νοοτροπιών είναι ο σύνδεσμος που αποκαθίσταται ανάμεσα σε έναν εργοδότη και ένα εργαζόμενο μέσα στο σπίτι, καθώς επίσης και ένα, ότι είναι περισσότερο μάλλον ένα σύνδεσμο συνεργασίας και όχι υποταγής. πρόκειται για κάτι διαφορετικό από το management που βλέπουμε σε μια επιχείρηση και βεβαίως εκεί είναι πολύ σημαντική η ανθρώπινη προστιθέμενη αξία και πολύ περίπλοκη. Αυτά φαίνονται από ορισμένες έρευνες και ανοίγονται εδώ κάποιες προοπτικές. Ένα από τα κύρια διακυβεύματα εδώ είναι και ο επαγγελματισμός. Προωθούμε δηλαδή τα προσόντα για να αναγνωριστούν ως επαγγέλματα οι οικιακές βοηθοί και οι γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά. Έχουμε δημιουργήσει επίσης μια ομάδα κοινωνικής προστασίας, ΙΡΣΕΜ, που φροντίζει ιδίως την κοινωνική στήριξη των οικιακών βοηθών και των ανθρώπων που φροντίζουν δικαιωμένα άτομα και παιδιά, για να έχουν την επιλογή οι οικογένειες να μπορούν να προσλαμβάνουν πρόσωπα δηλαδή για τις φροντίδες αυτές να βελτιωθούν οι συνθήκες, να ευαισθητοποιηθεί και να γίνει πιο υπεύθυνος εργοδότης, που είναι απαραίτητη από την πλευρά του εργοδότη, η ανάληψη της ευθύνη δηλαδή. Από το 2007 το IFPM οργανώνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο τις δραστηριότητες αυτές. Είναι ένας φορέας σήμερα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το λόγο αυτό που μπορούμε και συμμετέχουμε και στις δικές σας εργασίες σήμερα. Έχουμε απαντήσει και σε ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα και ένα που ολοκληρώνεται στο Παρίσι τις επόμενες εβδομάδες, Care Plus λέγεται αυτό, για ανθρώπους ηλικιωμένους και αυτούς που τους φροντίζουν στα σπίτια τους. Για να ολοκληρώσω θα έλεγα ότι οι μισθωτοί που εργάζονται σε καλές συνθήκες εργασίας, που κάνουν μια δουλειά μέσα σε σωστές περιστάσεις, προσφέρουν μια φροντίδα ποιότητας για την φροντίδα ανθρώπων που θεωρούνται εξαρτώμενοι, είτε πρόκειται δηλαδή για μικρά παιδιά, είτε πρόκειται για άρρωστους ηλικιωμένους. Είναι πολύ ουσιαστικό λοιπόν να γίνουν πραγματικοί επαγγελματίε οι άνθρωποι που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβετε υπόψη στην επόμενη θητεία σα, στην θητεία σα που αρχίζει δηλαδή, και να βοηθήσετε να προωθηθούν τα θέματα αυτά, γιατί και τα νοικοκυριά και οι οικογένειε έχουν και νέους ρόλους να παίξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο, μας έδωσαν πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε ένα τελευταίο μιλητή που θα μας μιλήσει για δύο-τρία λεπτά. Κέστιν Χάρβαλτ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδικάτων για τον Ρωτικό Τουρισμό και είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους που διοργανώσατε αυτή την εκδήλωση σήμερα και που μας ε, καλέσατε και μας δίνετε και το λόγο. Κάστιν Χούβερ, λέγομαι, εργάζομαι από τη μία συνομοσπονδία συνδικάτων της Ευρώπης, εκπροσωπώ και που εργάζονται στην γεωργία, στην βιομηχανία ε, τροφίμων, στον τομέα ξενοδοχείων, τουρισμού, αλλά εκπροσωπούμε και τους οικιακές βοηθούς, διότι τα περισσότερα εθνικά συνδικάτα στα οποία συμμετέχουν ε, οι εργαζόμενοι, είναι μέλλον της, μέλη της Συνομοσπονδίας. Γι' αυτό το θέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί με την Κάβε Πάρκερ από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οικιακών Βοηθών, που ξεκινά να δημιουργεί ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις οικιακές βοηθούς ε, μαζί με μας. Όπως είπα λοιπόν, τα μέλη μας Στη διάσκεψη συμμετείχαν ενεργά το 2011, οπότε και συνήφθηκε η 189 σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τους οικιακές βοηθούς. Πρώτο βήμα, χρειάζεται και επικύρωση βέβαια και εφαρμογή βέβαια της είναι λόγω συμβάσεως. Ε, ολοκληρώθηκε μια μελέτη περί βιομηχανικών σχέσεων στον τομέα αυτό Θέλαμε σαφή εικόνα του τομέα. Πώς οργανώνονται στη συνδικάτα και εκεί βοηθεί. βοηθή. Τι γίνεται με τις οργανώσεις εργοδοτών. Συλλογικές συμβάσεις στην Ευρώπη. Πώς ρυθμίζεται το τομέας. Είναι σημαντικό αυτό. Θέλουμε να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και εκεί βοηθεί. Κάτι πολύ δύσκολο που είπαν και οι προλαλήσαντες. Ο τομέας λειτουργεί βασικά ανεπίσημα και άτυπα μας ενδιαφέρουν, ε, θα μοιραστούμε τα πορίσματα της μελέτης μαζί σας. Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Σε κάποια κράτη-μέλη ε, ρυθμίζονται το τομέα, έχουμε κοινωνικό διάλογο και συλλογικές συμβάσεις. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όμως. Και στηρίζω αυτό που είπε η κυρία Λεβό. Πρέπει να συνεργαστούμε. Και οι εργοδότες και τα συνδικάτα να δημιουργηθεί περισσότερος κοινωνικός διάλογος. Μπορούμε να βασιστούμε στην αποκομιστήσα εμπειρία κάποιων κρατών μελών. Κοινός στόχος είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική κάλυψη για τους εργαζομένους στον τομέα, επαγγελματισμό, αναγνώριση και ρύθμιση νομική του θέματος. Καλούμε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κάνουν περισσότερα πραγματικά να ενθαρρύνονται τα κάτι μελη συνεχώς να κυρώσουν τη σύμβαση του Διεθνού Οργανισμού Εργασίας και να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία. Διότι τέσσερα χρόνια και ακόμα δεν, πέρασαν και δεν προχωρήσαν πολύ. Άλλο θέμα. Ζητούμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναθεωρήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να μην υπάρχει διάκριση κατά των οικιακών ε, βοηθών. Να μην αποκλείονται από κάποια δικαιώματα όπως η οδηγία για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Αποκλείονται από αυτήν ακόμα και εκεί η βοηθή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που έθεσε το θέμα αυτό της φροντίδας των οικιακών βοηθών. Ε, προσβλέπουμε να μάθουμε περισσότερα για την έκθεση. Η κυρία Κούνεβα θα συντάξει αυτή την έκθεση. Με τα χαράς να συμβάλλουμε κι εμείς, να δώσουμε από την εμπειρία μας Στι στις εργασίε εργασίες που θα γίνουν για το τομέα των οικιακών βοηθών. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος, ευχαριστώ όλους που πήραν το λόγο. Οπότε θα ακούσουμε και τα μέλη. Η κυρία Μορβάη έχει ζητήσει το λόγο και παρακαλώ μπορείτε να μιλήσετε μέσα σε δύο λεπτά. Θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ, λέει κυρία Μορβάη. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα από ό,τι κατάλαβα που και αυτό είναι διάκριση. Μιλώντας για διάκριση, ο τομέας της οικιακής εργασίας των οικιακών βοηθών στην Ευρώπη είναι μεγάλος τομέας διακρίσεων. Ε, η διάκριση με βάση το φύλλο αναφέρθηκε τους ομιλητές, προφανή διάκριση, αλλά η όλη ιδέα ότι η διάκριση ίσως να λήξει από τη στιγμή που Γερμανός, Γάλλος, Βρετανός ή Βρετανή, άντρας ή γυναίκα θα έχουν τις ίδιες πιθανότητες να καθαρίσουν τις τουαλέτες ενός Ούγκρου, ενός Ρουμάνου, ενός Ουγγρικού Ρωμανικού ε, νοικοκυριού και τούμπαλιν, τότε θα λήξει η διάκριση. Ή Γάλλος, οι Γερμανός, ή Βρετανός άντρας ή γυναίκα να αλλάξουν τις σύστηση να να καθαρισουν τις τουαλετες ενος ουγκρου ενος ρουμανου ενος ουγγρικου μωρών γερμανος η βρετανος αντας η γυναικα να αλλαξουν τις πανες μωρων η αναπήρων ή ηλικιωμένων στην Ουγγαρία ή στη Ρουμανία όπως και το αντίστροφο. Και θα πρέπει και αυτό το ευαίσθητο θέμα να το θίξουμε. Η ΔΕΜΗ, η νέα έκθεση αυτή, δεν θα είναι τόσο πολύτιμη όσο θα έπρεπε. Είναι θεμελιώδες θέμα δικαιοσύνης. Οι μετανάστες από τις ούτε αποκαλούμενες ε, χώρες του δευτέρας κατηγορίας και κυρίως άνθρωποι, γυναίκες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσης που είναι στη δεύτερη κατηγορία πολύ συχνά αυτοί αφήνουν τις οικογένειες τους πίσω, τις κοινότητες τους πίσω, τις πατρίδες τους πίσω για να πάνε σε πλουσιότερο κόσμο, τον κόσμο της πρώτης κατηγορίας και να ασχοληθούν με τις εργασίες αυτές. Πολύ συχνά είναι ε, ε, γυναίκες που έχουν επιτυχία κλπ. Αυτή η έκθεση λοιπόν θα πρέπει να εστιαστεί επ' αυτού. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να ρωτήσω όλους τους ομιλητές που πήγαν το λόγο τι είδους έρευνα έχει γίνει όσον αφορά αυτού του είδους την αδικία. Μα άλλα λόγια. Κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νέα κράτη τη μελη πρώην κομμουνιστικές χώρες. Οι γυναίκες από εκεί να ασχολούνται με κακή εργασία και να φροντίζουν υπηκόους χωρών πρώτης κατηγορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του δυτικού κόσμου του ΣΥΠΗΝ. Άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποιεί και καταχράτε το σύστημα ε, στα, στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης των εργαζόμενων στην Ευρώπη. Είναι πολύ παράξενο. Που αυτό είναι το επακόλουθο της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων. Δηλαδή φτωχές γυναίκες πάνε να καθαρίζουν τους τουαλέτες των πλουσίων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπήκαμε γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Εγώ θα μιλήσω ισπανικά. Σας ευχαριστώ. Χαιρετίζω τι εργασίε που κάνουμε για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι μια φορά και για πάντα θα πρέπει το θέμα αυτό να το θέσουμε επιτάπητο να το συζητήσουμε, διότι συζητούμε για τι ελλείψει που υπάρχουν ε, στο, στην ήπειρο εφημερία στην οποία ζούμε και αυτέ οι ελλείψει είναι ελλείψει από τι οποίε υποφέρουν οι εργαζόμενοι, εργαζόμενε κυρίω που δεν έχουν κανένα αναγνωρισμένο δικαίωμα. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε η εκπρόσωπος της Διεθνής Οργάνωσης Υγείας για τις ε, χώρες τις πιο ανεπτυγμένες στις οποίες ε, εργάζονται οι περισσότερες αυτές εργαζόμενες ε, αδήλωτες, χωρίς κανένα δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει επί της ουσίας να γίνει συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό συστημικό σφάλμα των συστημάτων. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε τέτοιες συζητήσει. Έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι ενδιαφέρουν τους πάντες και θα ήθελα απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο κανένα κανονιστικό ε, πλαίσιο που το οποίο θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε και σε άλλες χώρες. Σίγουρα στη χώρα της Ισπανία δεν υπάρχει, αλλά ισώ υπάρχουν άλλε χώρε, στι οποίε υπάρχει ένα νόμιμο νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να μα βοηθήσει και να μπορέσουμε το σύστημα αυτό, το πλαίσιο αυτό να το εξαγάγουμε σε άλλε χώρε. Δεύτερη ερώτηση προ την εκπρόσωπο τη Διεθνής Χρονιά εργασία. Τι είδου ε, δυσκολίε αντιμετωπίζετε με την επικύρωση, τι είδου ε, δυσκολίε υπάρχουν. Υπάρχει κάτι το οποίο αφορά ένα συγκεκριμένο μέρο τη σύμβαση. μπορείτε να το αναφέρετε για να δούμε κατά πόσον μπορούμε και να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Τρίτη ερώτηση, ίσως κάτι ε, το πιο περιορισμένο ενδιαφέροντος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις οικιακές βοηθούς στις πρεσβείες και στις ε, οικίες των ε, διπλωματικού σώματος στην Ευρώπη, διότι πρόκειται για άτομα τα οποία πραγματικά ζουν σε κατάσταση σκλαβιάς. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, διότι υπάρχει και θα, βγαίνει, θα πρέπει να δούμε περί τίνος πρόκειται, αν μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο στο φαινόμενο αυτό και να του δώσουμε περισσότερο φως. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα μέλη τα οποία θέλουν να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την δυνατότητα που μας δίνεται με την ακρόαση αυτή να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει και σημαντικό ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αλλά που άπτεται και πολλών άλλων θεμάτων σε άλλους τομείς που μας ε, είναι ιδιαίτερα προσφυλή σε εμά ε, τις γυναίκες στην Επιτροπή μας, αλλά και πολλούς άλλους ε, συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι υπάρχει πάντα η οπτική γωνία της απασχόλησης, του οικονομικού στοιχείου της ε, μετακίνησης των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέροντας ότι οι δύο μεγάλες δημογραφικές εξελίξεις, τα κλειδιά που εξηγούν τώρα τελευταία ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε οικιακές βοηθούς όλο και περισσότερο στα σπίτια μας, εξαιτίας όπως ελέγχθη εν μέρη της γύρας του πληθυσμού και δεύτερον διότι υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασία και εδώ έχουμε να κάνουμε με σημαντικά γεγονότα και τάσεις οι οποίες είναι κοινέ για τις περισσότερες χώρες. Είναι λοιπόν δική μας θέμα αρμοδιότητας, δική, θέμα δικής μας αρμοδιότητας να κάνουμε μετά από την διάγνωση για το πώς έχει η κατάσταση προτάσεις ώστε να μπορέσει το θέμα αυτό ευρωπαϊκά να βελτιωθεί και να συντείνουμε προς προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε το τι ακριβώς γίνεται και σωστή είναι εργασία και η τοποθέτηση της κυρίας Κούνεβα. Θα πρέπει να δούμε ποιες συνθήκες εργάζονται αυτοί οι εργαζόμενες. Αδήλωτες. και σφαιρικά να δούμε πώς συμπεριφερόμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση. Θα πρέπει να βγάλουμε από αυτή την φαιά ζώνη της ε, μη νομιμότητας ε, αυτής της εργαζόμενης, να το αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και να πούμε ότι πρόκειται για μια εργασία η οποία ε, θα πρέπει να έχει και να ειδωθεί ως μια, ένα επάγγελμα Δεδομένου ότι πρέπει κανείς να έχει επαγγελματικά προσόντα, προσόντα τα οποία θα πρέπει να τα ε, συζητήσουμε και με τους ε, εκπρόσωπους εργαζομένων και εργοδοτών. Σε πρώτη φάση θα πρέπει λοιπόν να βγουν από την αφάνεια και την παρανομία αυτοί οι εργαζόμενοι ώστε να επιτευχθεί πρόοδος. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να συγκεράσουμε την ε, οικιακή εργασία με την πρόοδο την κοινωνική. Πρόκειται για, μια, για ένα στίχημα μεγάλο, διότι βλέπουμε ότι πρόκειται για μια πρακτική η οποία είναι πρακτική ίσως όχι μόνο ετών και δεκατιών αλλά και ενώνων σε κάποιες χώρες. Και όπως είπε και η Γαλλίδα συνάδελφος, στην Γαλλία άλλαξαν τα πράγματα αλλά υπάρχει και σημασιολογική ε, ε, σημασία στο όλο πρόβλημα και γρήγορα πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες για να αλλάξουν τα πράγματα και η πρακτική που ακολουθείται σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Το θέμα λοιπόν αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το συνδέσουμε ε, με, απευθείας με την κοινωνική πρόοδο την οποία θέλουμε να επιτελέσουμε στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το σχολείο μου. Δεν ήθελα να κάνω ερωτήσεις, αλλά επιμένω θα πρέπει να προσπαθήσουμε το θέμα αυτό να το συνδυάσουμε και πάλι με την κοινωνική πρόοδο, με την πρόοδο κάθε ανθρωπίνου όντως στις κοινωνίες μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα αυτά προβλήματα και τις προκλήσεις που έχουμε και πάλι επαναλαμβάνω το θέμα της γύρανσης και θα πρέπει όντως η εργασία που γίνεται στον τομέα αυτό να γίνεται νόμιμα και με όλες τις κοινωνικές παροχές που πρέπει. Και βεβαίως έχουμε να κάνουμε με άτομα τα οποία φροντίζουν τα παιδιά, του ηλικιωμένου, τα άτομα τα εξαρτώμετα, τα άτομα με αναπηρίες που ε, πρέπει να έχουν και κάποια επαγγελματικά προσόντα. Και να το λέει και η ψυχούλα τους αν θέλετε για να ασχολούνται συνέχεια με τα θέματα αυτά που είναι τόσο σημαντικά. Ευχαριστώ. Ε, χαιρετίζω την εργασία που συλλογικά θα επιτελέσουμε για να πετύχουμε το στόχο μας αυτό. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλα μέλη που επιθυμούν να λάβουν το λόγο, θα ζητούσα από καθέναν από τους τέσσερις φιλοξενούμενους μας να πούν μερικά λόγια εν κατακλείδη. Φοβούμαι ότι θα πρέπει να περιοριστούμε χρονικά στα τρία λεπτά ο καθένας, διότι πρέπει να τελειώσουμε εγκαίρως. Ο κύριος Καπαρίτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, την μετακίνηση, την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη, η έρευνά μας που έγινε πρόσφατα για την εργατική κινητικότητα στην Ευρώπη δείχνει ότι, είναι αρκετά μέτρη ρυθμή αριθμητικά 0,03% διασυναριακής ε, κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών. Μπορούμε πάντα να εξετάσουμε τα στοιχεία. Σχετικά όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μετακίνηση από ανατολικά προς το δυτικά κυριαρχεί το και οι βασικές κινήσεις νότου-βορρά. Υπάρχει, είναι πιο έντονη η μετακίνηση ανατολικά προς δυτικά από ότι από νότον προς βορρά. Και η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι, αυτές, ε, είναι η πόλη έλξης για τους μετανάστες. Και κάτι άλλο. Καμιά φορά σκεφτόμαστε υπηκότητα. Εξετάσαμε όμως και συνθήκες εργασίας κατά το παρελθόν ανθρώπων που προέρχονται από το εξωτερικό. Εργαζομένους δεύτερης τρίτης γενιάς, α, που γεννήθηκαν σε μια χώρα, αλλά η καταγωγή τους δεν είναι από αυτή τη χώρα. Οι γονείς τους δεν κατάγονται από τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν αυτοί. Άρα μιλάμε για εργαζομένους δεύτερης ή τρίτης γενιάς και τα στοιχεία δείχνουν ότι και αυτή ίσως να είναι αντικείμενο διάκρισης και ίσως να εργάζονται σαν οικιακή βοηθή ε, στις οικοδομές κλπ. Όμως, απλευράς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος από το εξή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, δημογραφικές εξελίξεις κλπ. Και τομεακές προσαρμογές που βλέπουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία. Βλέπουμε ότι ο τομέας αυτός θα αυξηθεί στο μέλλον. Δοθέντος και του άτυπου χαρακτήρα του, αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Θα αυξηθεί σαν τομέας. Δεδομένο αυτό. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσουμε ότι οι συνθήκες για τις νέες θέσει εργασία θα είναι καλές, να είναι ποιοτικέ θέσει. Αξιοπρεπή αμοιβή, αξιοπρεπέ συνθήκε εξασφαλίζεται υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Σας είπα το πρωί ότι όσον αφορά τους οικιακούς βοηθούς που μένουν στο σπίτι υπάρχουν κίνδυνοι που είναι πάνω από το μέσο όρο και θα πρέπει να το καλύπτει η νομοθεσία όσον αφορά τις καλές πρακτικές. Ο Ισπανός συνάδελφος το έθεσε. ρίξε μια ματιά στην έκθεση. Έχω καπεντίγραφα εκεί. Που θέλουμε καλύτερε θέσει εργασία όσον αφορά την παροχή ε, περίθαλψη στο σπίτι. Έχουμε πολλά καλά παραδείγματα, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά. Πώ μπορεί κανεί να πετύχει καλύτερε θέσει εργασία και περισσότερο περισσότερες σε αυτό το τομέα. Και πολλά από αυτά τα ε, παραδείγματα μπορούν να ε, ληφθούν υπόψη και στην κατοίκον φροντίδα. Πολλά, πολλοί από του εργαζομένου δεν συμμετέχουν, δεν είναι μέλη συνδικάτων, η οργάνωσή του δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που μπορούν να του βοηθήσουν να δοθεί, να αναγνωριστούν τα προσόντα τους, ε, η εκπαίδευσή τους ε, και μέσω αυτού να βελτιωθούν οι διαθέσιμε θέσει εργασία και να αναβαθμιστούν και στο μέλλον. Δεν θέλουμε απλώς περισσότερες θέσεις εργασίας, θέλουμε και καλύτερες θέσεις εργασίας. Να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εργασίας των θέσεων που θα δημιουργηθούν στο μέλλον και σε αυτόν τον τομέα και σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Κύριε Ψημένε. Ε, ε, έχουμε περάσει περίπου 25 χρόνια στη χώρα μας μελετώντας την οικιακή εργασία και άλλες μορφές εργασίας ανάμεσα σε αυτήν είναι και η εργασία σε ε, μεταναστριών σε ε, υπηρεσίες ε, που παρέχονται παράνομα ή νόμιμα και ονομάζονται σεξουαλικές υπηρεσίες. Έχω την εντύπωση ότι τα διλήμματα τα οποία διακυβεύονται αυτή τη στιγμή είναι βασικά τρία. Το ένα είναι η κοινωνική προστασία εργαζομένων σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να είναι άτυπο ή τυπικό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε κίνητρα και πώς θα δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι ώστε οι μετανάστες οικιακές εργάτριες να μπορέσουν να δηλώσουν το επάγγελμά τους στις αρχές και στην κοινωνική πρόνοια και να μπορέσουν να έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτό για να γίνει βεβαίως απαιτεί να προσέξουμε πάρα πολύ ποιες παραμέτρους επηρεάζουν την είσοδο και την τον εγκλωβισμό των οικιακών εργατριών μέσα στην άτυπη εργασία. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο επίσης πρέπει να προσέξουμε είναι η κινητικότητα. Μιλάμε για την επαγγελματικοποίηση της οικιακής εργασίας. Κάποιοι ε, ε, ε, συνάδελφοι και αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου θεωρούν ότι αυτός θα είναι ο δρόμος για να λύσουμε τα προβλήματα της οικιακής εργασίας. Θεωρώ ότι το βασικό το πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε διαμορφώσει μια Ευρώπη τριών, τεσσάρων ή πέντε ταχυτήτων. Πολύ σωστά προηγουμένως αναφέρθηκε ότι συγκεκριμένες γυναίκες από συγκεκριμένες χώρες με συγκεκριμένα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά καθαρίζουν τα σπίτια μας. Αυτό το φαινόμενο δεν ονομάζεται ούτε επαγγελματικοποίηση ούτε τίποτε άλλο. Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο λάθος εάν δημιουργήσουμε μια βικτοριανή, νέο βικτοριανή εποχή ότι όπου το μόνο το οποίο θα λείπει στην Ευρώπη είναι σχολές οικιακών εργατριών. Σε αυτό εγώ προσωπικά και οι μελέτες μας οδηγούν ότι πρέπει να είμαστε αντίθετοι. Το τρίτο θέμα το οποίο επίσης νομίζω ότι πολλές φορές μας διαφεύγει είναι ότι οι οικιακέ αυτές εργάτριες έχουν οικογένειες. Η οικογενειακή επανέναση στην Ευρώπη είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να μην το ανοίξουμε ως μία ατζέντα. Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον κόσμο με τις καλύτερες συνθήκες που να αισθάνεται ότι αναπτύσσεται ο εαυτός του μακριά και ξέχωρα από την οικογένειά του και από τη δυνατότητα ανάπτυξης οικογενειακών σχέσεων. Ιδάλλως Πολύ φοβάμαι ότι τα 4 ή 7 εκατομμύρια οικιακών εργατριών θα πρέπει να μην ονομάζονται οικιακές εργάτριες, αλλά χωρίς οικογένειε οικογένειές να ονομάζονται οικιακοί σκλάβοι. Εάν η Ευρώπη έχει μία δυνατότητα είναι να δει ότι προσκρούει κάθε ανάπτυξη της οικιακής εργασίας σε τρεις βασικές ελευθερίες. Προστασία, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη και οικογενειακές σχέσεις. Αυτά είναι τα τρία, οι τρεις πυλώνες κοινωνικής πολιτικής που θα πρέπει η Ευρώπη άμεσα να κοιτάξει και να μπορέσει να, για να μπορέσει να υπάρξει μια καλύτερη συνθήκη στις εργαζόμενες μετανάστριες. Τέλος θέλω να πω κάτι. η επικύρωση της σύμβασης και των συμβάσεων. Ξέρετε κάτι, εάν κάθομαι και σκέπτομαι πόσο σημαντική είναι μια επικύρωση μια σύμβαση. Αλλά θα ήθελα να ξέρω σε ποιες χώρες οι συμβάσεις αυτές και σε, ε, σε ποια ιδιωτικά νοικοκυριά θα έχουν καμία ισχύ. Τη στιγμή που περισσότερο αυτό που μας απασχολεί είναι να μην πάνε οι γυναίκες μέσα στα σπίτια, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξεις ουσιαστικά την ε, ε, οικιακή εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος, κυρία Κουλτάη. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση, για την μετανάστευση. Δυστυχώς δεν έχω τα συγκεκριμένα στοιχεία που ζητείτε. Αυτό που γνωρίζουμε ως Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι ότι υπάρχει, για παράδειγμα, η γλώσσα είναι πολύ σημαντική. Στην Ισπανία οι περισσότερες οικιακές εργάτριες έρχονται από τη Λατινική Αμερική. Στη Γερμανία οι περισσότερες έρχονται, ε, στη Γαλλία, συγγνώμη, στη Γαλλία, έρχονται από τις χώρες Μαγκρέμπ. Ε, η κυρία Μορβάη, νομίζουμε χωρίς μικρόφωνο ότι λέει γιατί δεν πάνε και ανάποδα. Δεν έχω βεβαίω απάντηση στην ερώτηση αυτή, αυτό είπα και από την αρχή τη απάντησή μου. Αυτό που βλέπουμε, δηλαδή γιατί δεν πάνε στην άλλη κατεύθυνση, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί δεν πάνε από τη Γερμανία, δηλαδή να καθαρίζουν τουαλέτε στην Ουγγαρία, αυτό δεν το ξέρω δεύτερο του Ισπανού συναδέλφου σας. Ποια είναι τα εμπόδια και γιατί δεν, δεν, δεν κυρώνουν περισσότερες χώρες την σύμβαση. Δεν έχω και εκεί όλες τις απαντήσεις, αλλά προτιθέμεθα να κάνουμε ένα εργαστήριο μαζί με προσώπηση των χωρών μελών για να δούμε. Υπάρχει ωστόσο σαφώς ένα θέμα προτεραιότητας τα επιχειρήματα υπέρ ή μάλλον η πίεση για μια κύρωση δεν είναι πολύ ισχυρή, διότι δεν είναι οργανωμένε οι οικιακέ εργάτριε. Δεύτερο, σε πολλέ χώρε μέλη δεν υπάρχει παραδοσιακά κάποια τέτοια στάση για επαγγελματικοποίηση των ε, ε, οικιακών εργατριών και ίσω γι' αυτό να διστάζουν ορισμένε χώρε μέλη. Και τώρα επίση, σε ορισμένε χώρε μέλη υπάρχει μια έλλειψη αναγνώριση τη κατάσταση των οικιακών εργατριών. δεν αναγνωρίζουν απαραίτητα τα θέματα που μπαίνουν από την εργασία αυτή. Δεν είναι στην ατζέντα τους ας πούμε. Βέβαια ίσως υπάρχουν και κάποια τεχνικά εμπόδια τα οποία δεν τα ξέρω ακόμη και θα τα βρούμε ίσως με το εργαστήριο που θα κάνουμε. Και θα σας ενημερώσω τότε. Σας ευχαριστώ. Και τελευταία η κυρία Λεβό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εγώ εκπροσωπώ την ε, ε, κοινωνία των πολιτών και εδώ επευθύνομαι σε πολιτικούς. Ο καθένας στη θέση του λοιπόν και υπάρχουν θέματα που δεν μπορώ να απαντήσω είναι τις μου. Θα ήθελα να πω παρόλα αυτά ότι την άποψή μου δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα μελετήσουμε και εσείς να ασχοληθείτε δεδομένου ότι είστε πολιτικά υπεύθυνοι. Πρώτα απ' όλα, να αγωνιστούμε κατά. Πολλοί λέγουν πολύ σωστά πράγματα. Κατά της παρανομίας, κατά αυτού του... Ε, χαρακτήρα το ότι δεν φαίνεται πουθενά αυτή την... Ε, δεν πουθενά αυτοί οι άνθρωποι κατά της νομοθεσία αν δεν το βοηθάει. Πιστεύω λοιπόν ότι και εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι ώστε να δώσετε μία προσθέμενη αξία στην αναγνώριση της εργασίας, των επαγγελμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων που μπορούν να δημιουργήσουν νέα επαγγέλματα, νέε αρμοδιότητες, νέα προσόντα. Δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που υπάρχουν για τη σημερινή ζωή των ανθρώπων όταν μιλούμε μόνο για την οικιακή εργασία και αναφέρομενται μόνο στους μετανάστες. Το 20% τη Γαλλία των εργασιών σήμερα εκτελούνται από μετανάστες ενδοκοινοτικούς και εξοκοινοτικούς. Πολλές όμως θέσεις απασχόληση ε, είναι θέσεις τις οποίες κατέχουν οι νέοι μας σήμερα και έχουν έναν ανθρωπιστικό σημαντικό χαρακτήρα, κυρίως όταν πρόκειται για άτομα τα οποία πρέπει να φροντίσουν άτομα τα οποία δεν έχουν, ε, πρέπει, άτομα τα οποία έχουν προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ανοίξουμε και στον κοινωνικό τομέα νέες καινοτόμους ε, και οδούς. Πρέπει όντως να ε, καταπολεμήσουμε αυτά τα οποία αναφέρεται. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι η Γαλλία, και το λέω με μεγάλη ταπεινοφροσύνη, ότι πρόκειται για μια χώρα που έχει τις βέλτιστες ε, πρακτικές, διότι θέλει μέσω των συλλογικών συμβάσεων να διασφαλίσει όλους τους εργαζόμενους. Και αν υπήρχε κάτι το παραφερέ σε όλες τις χώρες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Δεύτερον, πώς μπορούμε σε αυτά τα οποία έχουμε στη θεωρία να δώσουμε στην πράξη αξία. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι σωστά και πρέπει να τα βελτιώσουμε. Ούτω ή άλλω κανένα κράτο δεν έχει του πόρου που χρειάζεται, του δημόσιου πόρου για να βελτιώσει την κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν σύμπραξη όλων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τι τέσσερι ομιλητέ και να δώσω τώρα στην εισηγήτρια την κυρία Κούνεβα το λόγο για τα συμπεράσματα και να μας πείτε και λίγο τι πραγματεύεται η δική σας έκθεση. Ευχαριστώ πολύ όλους όσου ήρθαν σήμερα εδώ για να μας δώσουν τα φώτα τους και να μοιραστούν τις γνώσεις τους με μας. Ε, η συνεργασία φέρνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Η... Στηρίζουμε σε όλες τις καλές ιδέες και την διάθεση των συνάδελφων μου για να προσφέρουμε στους οικιακούς εργαζόμενους την αξιοπρέπεια που τους αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you all very... Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε, πέμπτη μάλιστα, ημέρα πέμπτη της εβδομάδας. Βρήκα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον σε συζήτηση και μας πρόσφερε όπως είπα τροφή για σκέψη. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε στο σημαντικό αυτό θέμα. Σας ευχαριστώ.